Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σα καλωσορίσω όλους και όσους ε, συμμετέχουν αυτοπροσώπως και εξ αποστάσεως και τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών που ενδεχομένω παρακολουθούν τη Σύνοδο τη Ολομέλειας. Πρώτα θα ήθελα να κάνω μία ανακοίνωση για τη σύνθεση των επιτροπών μετά τη σύσταση των επιτροπών αναγγέλθηκαν οι διορισμοί στις επιτροπές βάσει του άρθρου 209. Οι ειδικέ επιτροπές είναι ακόλουθες. Ειδική Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη, Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, Επιτροπή για τις ξένες παρεμβάσεις και την παραπληροφόρηση, τα fake news, Επιτροπή για τη φορολογία και επιτροπή για τη μεταφορά ζώων. Η σύνθεση των νέων επιτροπών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η επόμενη ανακοίνωση η ανακοίνωση για την έναρξη διοργανικών συνομιλιών και διαπραγματεύσεων ε, από διάφορες επιτροπές. Πολλές επιτροπές αποφάσισαν την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων, όπως ε, ανακοινώθηκε ε, στις 8 Ιουλίου κατά την έναρξη της Συνόδου της Ολομέλειας. Δεν υπευλήσαν αντιρρήσεις, οπότε μπορούν οι Αντίστοιχε επιτροπέ να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσει. Πριν όμως περάσουμε στην ημερήσια διάταξη, να σας ανακοινώσω τα αποτελέσματα της ε, χθεσινής ε, τρίτη ψηφοφορία. Στα αγγλικά, έκθεση Kovarik για τι ημερομηνίε μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή εξαιτία τη έξαρση τη κρίση ε, τη πανδημία COVID-19. Εγκρίνεται. Έκθεση Command, Οικονομικέ δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2019 εγκρίνεται. Έκθεση ECHOT, Ετήσια Έκθεση 2018 για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εγκρίνεται. Έκθεση ΚΟΥΧ για την καταπολέμηση τη απάτη. Ετήσια Έκθεση 2018 εγκρίνεται. Κοινό ψήφισμα τριών ομάδων. Ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Εγκρίνεται ψήφισμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 για τις ε, δραστικές ε, ουσίες. Τροπολογία 1 εγκρίνεται. Τροπολογία 2 εγκρίνεται. Τροπολογία 3 εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ΤΑΦ απορρίπτεται. Ψήφισμα της Επιτροπής Βιομηχανίας ε, για την ε, μεταρρύθμιση των ε, κατευθυντηρίων γραμμών για τι υποδομέ διαδικτυακών δικτύων μεταφορών. Ε, πρώτο τμήμα τροπολογία 1 απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα τροπολογία 1 απορρίπτεται. Τροπολογία 5 απορρίπτεται. Τροπολογία 6 απορρίπτεται. Τροπολογία 7 απορρίπτεται. Τροπολογία 8 απορρίπτεται. Τροπολογία 9 απορρίπτεται. Παράγραφος 3. Αρχικό κείμενο. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4. Πρώτο τμήμα. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Δεύτερο τμήμα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Απορρίπτεται. Και τροπολογία 4. Επίσης απορρίπτεται. Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Νέα Ζηλανδία για την ε, ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων για την καταπολέμηση σοβαρού εγκλήματο και τρομοκρατία. Τροπολογία 2. Απορρίπτεται. Θεωρώντα 13. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη F. Πρώτο τμήμα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Εγκρίνεται. Και τρίτο τμήμα επίση εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη H. Αρχικό κείμενο. Καταπίπτει. Ψήφισμα τη Επιτροπή Περιβάλλοντο για τη στρατηγική για τι χημικέ ουσίες ε, εν ώψη τη βιωσιμότητα. Τροπολογία 1. Απορρίπτεται. Παράγραφο 21. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Τμήμα 2 της 21 εγκρίνεται. Παράγραφος 22. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα επίσης εγκρίνεται. Παράγραφος 23. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Και δεύτερο τμήμα εγκρίνεται ομοίως. Παράγραφο 41. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Απορρίπτεται. Παράγραφος 81. Εγκρίνεται. Παράγραφος 82. Πρώτο τμήμα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Το πρώτο τμήμα εγκρίθηκε, το δεύτερο απορρίφθηκε. Τροπολογία 5. Απορρίπτεται. Παράγραφος 86. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Απορρίπτεται. Παράγραφος 116. Εγκρίνεται. Θα κάνουμε τώρα μία σύντομη διακοπή, λιγόλεπτη, και η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 9 και 4. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Θα ε, προχωρήσουμε ε, στη συζήτηση. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα λάβει το λόγο ένας ε, ομιλητής από κάθε πολιτική ομάδα και δεν θα έχουμε διαδικασία αυθόρμητων τοποθετήσεων ΚΑΤΣΙΑΗ ούτε γαλάζιες κάρτες. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Επιτροπής για την εκδήλωση μνήμης ε, για τη Σερμπρένιτσα με τη συμπλήρωση 25 ετών. Ε, δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κύριο Βάρχελη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σήμερα θυμόμαστε μία από τις πιο σκοτεινές ημέρες της σύγχρονης ε, ευρωπαϊκής ιστορίας. Μία, ένα από τα πιο τραγικά εγκλήματα που διαπράχθη στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον Ιούλιο του 1995, πάνω από 8.372 μουσουλμάνοι άντρες και αγόρια σκόπιμα και συστηματικά δολοφονήθηκαν από τις, Βοσνι... από τις δυνάμεις της Βοσνίας στην περιοχή της Σεμπρενίτσα μια πόλη που θεωρούσαν αυτοί οι άνθρωποι ότι ήταν ασφαλής από τον πόλεμο που σοβούσε ε, στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Οι σωροί τους ρίχθησαν σε μαζικούς τάφους με το πρόσωπο προς το έδαφος και τα χέρια δεμένα. Τα τελευταία θύματα ετάφησαν με τιμές. Η σκέψη μας και η καρδιά μας είναι με αυτούς και με τους ε, επιζήσαντες, τους φίλους τους, ε, τις οικογένειές τους θυμόμαστε και τιμούμε ε, τα θύματα και απευθύνουμε τη συμπάθειά μας και τα συναισθήματά μας συμπαράσταση σε αυτούς που θρηνούν και ελπίζουμε να θεραπευθεί ο πόνος τους. Η Ευρώπη δεν έχει λησμονήσει αυτό που συνέβη στη Σερμπλενίτσα και την ευθύνη μας που δεν μπορέσαμε να εμποδίσουμε, δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε αυτή την γενοκτονία. Στη Σρεμπρενίτσα απέτυχε η Ευρώπη και αντιμετωπίζουμε το όνειδός μας. Πράγματι η γενοκτονία της Ρεμπερενίτσα παραμένει μια χαίουσα πληγή και η καρδιά της Ευρώπης εξακολουθεί να στοιχιώνεται από αυτό το γεγονός. Θυμόμαστε τις κοινέ ευθύνε που έχουμε για να αποφύγουμε την γενοκτονία, να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο ποτέ. Γι' αυτό έχουμε καθήκον να θυμόμαστε τη Σρεμπρενίτσα πάντα. Επίσης έχουμε καθήκον να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει λογοδοσία. Δικαιοσύνη θα πρέπει να αποδοθεί. Και όλοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τη σφαγή θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την συνέπεια, τις συνέπειες των πράξεών τους. Μετά από 25 χρόνια, τώρα είναι πιο επίγον από ποτέ να σταματήσει η ατιμορρησία για εκείνου που διαπράττουν εγκλήματα πολέμου, διέπραξαν εγκλήματα πολέμου. Η σφαγή τη Εμπερενίτσα αναγνωρίστηκε σαν πράξη γενοκτονία από δύο διεθνή δικαστήρια διαφορετικά, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην το 2004 και το διεθνέ Διεθνές Δικαστήριο το 2006. Αυτά είναι αποδεδειγμένα γεγονότα αυτά που συνέβη σε Σεμπρενίτσα. Πρέπει να γίνουν αποδεκτά. Οποιαδήποτε απόπειρα άρνησης, αναθωρητισμού είναι πράγματα απαράδεκτα. Οι πολιτικοί ηγέτες έχουν μεγάλη ευθύνη όσον αφορά το θέμα πρέπει να επιλέξουν την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τη συνεργασία πάνω από το φόβο και το μίσος, ούτω ώστε να ξεπεραστεί η ταγική κληρονομιά του παρελθόντο και να οικοδομηθεί λαμπρότερο και πιο ευημερές μέλλον για, το, για γενιές. Οι ηγέτες της περιοχής θα πρέπει να οικειοποιηθούν αυτό που συνέβη και να δώσουν το καλό παράδειγμα. Δεν υπάρχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ρητορική μίσους, και το να δοξάζονται εγκλήματα πολέμων, πολέμου από τις διάφορες πλευρές. Οι πολιτικοί ηγέτες θα πρέπει να προσπαθούν τους πολίτες, τους κυρίως τους νέους, να τους συναθρίζουν σε ένα κοινό όραμα για το μέλλον, να υπάρχει εμπιστοσύνη, αμοιβαία κατανόηση και να σέβονται όλοι τους άλλους. Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να συμβάλλει σε ένα τέτοιο μέλλον. Ε, είναι θεμελιώδη σημασία. Παίζει ζωτικό ρόλο στο να τροφοδοτεί δημοκρατική νοοτροπία να υπάρχει ανάμνηση των γεγονότων και στα Δυτικά Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη, κυρίως προς όφελος των νέων γενεών. Από όλου μας στην Ευρώπη εξαρτάται να μάθουμε τα μαθήματα από τη Σερμπερνίτσα. Παραβιάστηκαν εδώ και 25 χρόνια βία πολλές αξίες. Ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, Αυτές οι αξίες είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών που καταβάλλονται στη Βοσνία Ζεγοβίνη από τους πολίτες τους. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζουμε αυτές τις αξίες σε όλες μας τις σχέσεις με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Τον εφαρμόζουμε αποφάσει διεθνών δικαστηρίων και τον προωθούμε ένα περιβάλλον που οδηγεί σε συμφιλίωση. Αυτό θέλουμε για να ξεπεραστεί η κληρονομιά του πολέμου. Αυτά είναι βασικά στοιχεία για όλες τις χώρες της περιοχής, ώστε να προοδεύσουν και να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προωθήσουμε συμφιλίωση σε όλα τα επίπεδα να εξασφαλίσουμε μακροπρόθεσμα την καθημερινή ζωή αυτών των ανθρώπων. Κάθε πολίτη συνεπάγεται αποζημίωση στα θύματα του πολέμου, εκείνο που ήταν θύματα βασανιστήριων, βιασμών, να υποστηρίξουμε την επιστροφή των εκτοπιστέντων και των προσφύγων και να επιτρέψουν στι οικογένειε των αγνωμένων να τελικά να μπορέσουν να ξεπεράσουν τον πόνο του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίσει να υποστηρίζει τη Βοσνία Ζεγοβίνη, ώστε να προχωρήσει στο μονοπάτι προ την Ευρώπη, παγιώνοντα μια κοινωνία πλουραλισμού δικαιοσύνη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μέσω τη συνταξιακή διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθεί να συνοδεύει τα Δυτικά Βαλκάνια προ τη συμφιλίωση και περιφερειακή συνεργασία, ούτω ώστε να δημιουργηθεί ένα ευημερέ και ε, ειρηνικό μέλλον για όλου του λαού τη περιοχή. Το να παραδεχθούμε το παρελθόν θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Πράγματι, χωρίς τη συμφιλίωση δεν θα υπάρξει μακροπρόθεσμη ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στα Δυτικά Βαλκάνια. Γι' αυτό καλό τα Δυτικά Βαλκάνια να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, να επουλωθούν οι πληγές του παρελθόντος και να πετύχουμε μια κοινή Ευρώπη. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Σας ευχαριστώ. Ε, ο επόμενος ομιλητής από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Παύλο Ρανζέλ. Παρακαλώ. Never again. Ποτέ πια, ποτέ πια, ποτέ πια. Ποτέ ξανά, Πρόεδρε, Επίτροπε. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την κραυγή ε, αυτό το πελπισμένο μήνυμα σε όλους τους Βόσνιους πολίτες, ανεξαιρέτως, αδιακρίτως θρησκείας, πίστης, έθνους. Θα ήθελα όμως να το απευθύνω αυτό και σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που στο παρελθόν έζησαν τη φρίκη και την κόλαση της γενοκτονίας. Για να το πω καλύτερα σε όλη την ανθρωπότητα το απευθύνω. Η θυσία της Σερμπρένιτσα δεν είναι μόνο η τραγωδία για ε, ε, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είναι η ίδια η άρνηση της ανθρωπιάς. Όποτε και όπου επιτελείται γενοκτονία, σφαγή, μαζική και συστηματική θανάτωση αθώων, είναι η ίδια η άρνηση ε, της ανθρωπιάς, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εκεί είναι πάντα μια Σρεμπρένιτσα. Όλες οι γενοκτονίες, αλλά ιδιαίτερα εκείνη τη Σρεμπρένιτσα απαιτούν αλήθεια και δικαιοσύνη που είναι η πεμπτουσία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του σεβασμού. Η αλήθεια δεν είναι συμβατή με την άρνηση. Η δικαιοσύνη δεν συμφιλιώνεται με την ατιμορρησία. Εξ ονόματος των Ευρωπαίων πολιτών που εμείς εκπροσωπούμε θέλω να δείξουμε τη συντριβή μας και την βαθύτατη ντροπή μας απέναντι σε όλα τα θύματα της Ρεμπρένιτσα, σε όλους τους επιζώντες και τις οικογένειες και σε όλους τους Βοσνίους και τολμώ να πω και προς όλη την ανθρωπότητα. Κάποιοι ε, ε, ήταν υπεύθυνοι ε, για αυτή τη σφαγή, ε, αλλά ε, είναι αδικαιολόγητη και ασυγχώρητη η ολιγορία και η αδράνεια της Ευρώπης και των άλλων διεθνών θεσμών. Χωρίς τη δίψα για δικαιοσύνη των θυμάτων και των οικογενειών δεν νοείται συμφιλίωση. Υπάρχει όμως και ελπίδα για ένα μέλλον ε, με ευημερία και ειρήνη για όλη τη Βοσνία Ζεγοβίνη και όλους τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών το λόγο έχει ο κύριος Πίτσο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Με βαθύτατη λύπη και ιδιαίτερη κατάνοιξη προς τα θύματα ε, ε, της μεγαλύτερης ε, τραγωδίας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλούμε για τη γενοκτονία στην Σρεμπρένιτσα. Συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από την γενοκτονία αυτή, αλλά η μνήμη των απότροπων σκηνών βρίσκεται ακόμη ζωντανή μέσα μας. Πριν από πέντε χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ιδιαίτερο ψήφισμα για τη γενοκτονία στην ε, Σρεμπρένιτσα. Για όσου έχασαν του αγαπημένου του, βέβαια δεν υπάρχει παρηγοριά. Και όπω είναι σημαντικό να ταυτοποιηθούν τα λείψανα των θυμάτων, είναι σημαντικό να ταυτοποιηθούν και το έγκλημα και οι εγκληματίε. Τα δικαστήρια στη Χάγκη, Βοσνία Ερζεγοβίνη, στη Σερβία και την Κροατία καταδίκασαν ε, πάνω από 47 ε, κατηγορούμενους σε κάθριξη άνω των 700 ετών για συμμετοχή σε γενοκτονία που διεπράχθη στη Σρεμπρένιτσα. Ναι, το έγκλημα στη Σρεμπρένιτσα είναι γενοκτονία και έτσι θα πρέπει να το χαρακτηρίσουμε. Έχουμε τι αποφάσει, τι δικαστικέ του Διεθνού Δικαστηρίου για την πρώην Ιουκοσλαβία και του Διεθνού ε, Δικαστηρίου. Αλλά η πάροδο του χρόνου ενδύνει την υποχρέωσή μα να προστατεύσουμε τα θύματα από την προγραμματισμένη λύθη μέσω πολιτικών τεχνασμάτων, γιατί τέτοιε προσπάθειε γίνονται και θα γίνονται από την απονομή βραβείου Νόμπελ σε εκείνων που αρνούνται τη γενοκτονία, μέχρι παραπληροφόρηση ανερχιστρωμένη από διάφορα αυταρχικά καθεστώτα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο έγκλημα να θριαμβεύσει εκ των υστέρων. Αυτό οφείλουμε στα θύματα τη Ρεμπρένιτσα, αλλά και τη Όφτσερα και άλλων μεγάλων μαζικών εκτελέσεων που άφησαν το το, το ίχνος της του σχεδίου της Μεγάλης Σερβίας. Ε, Σίγουρα μόνο η πρόσπιση τη αλήθεια ανοίγει καλύτερο μέλο για τι επερχόμενε γέε. Ο πλούτο τη ε, Βοσνία Ερζεγοβίνη έγκυται στην πολυεθνωτική τη ε, ε, κουλτούρα, ε, στις, ε, στις πολλές θρησκείες, όλες οι θρησκείες και εθνότητες εκεί αξίζουν πλήρως σεβασμού. Και αυτό είναι το εχέγγυο ε, για το, το μέλλον της. Μια σαφή προοπτική της ε, Βοσίνης Ριζεγοβίνης για ένταξη το οφείλουμε στα θύματα της ε, Σρεμπρένιτσα αλλά και στους νέους που προσβλέπουν να ζήσουν σε μια ειρηνική και ευήμερη περιοχή. Και αυτό είναι σημαντική, σημαντικό αχέγιο για την πρόοδο της χώρας. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής εκ μέρους της ομάδας Renew είναι ο κύριος Φλέγκο. Παρακαλώ. Αξιότιμα κύριε Επιτροπέ, συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από το πιο αποτρόπαιο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 25 χρόνια πέρασαν από τη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα και κανένας δεν έχει δικαίωμα να αρνείται την γενοκτονία αυτή στη Σρεμπρένιτσα και να σχετικοποιεί τα γεγονότα. Και λυπάμαι πραγματικά ειλικρινά που δεν υπήρξε η πολιτική θούλης, βούληση και το θάρρος για ε, μια, ένα ψήφισμα για την ε, Σρεμπρένιτσα μετά τη συμπλήρωση 25 χρόνια από την τραγωδία. Και μάλιστα το ότι δεν στυλιτεύουμε τους εγκληματίες είναι μεγάλη αποτυχία της κοινωνίας μας. Μόνο η αλήθεια είναι το εχέγγυο για τα θύματα. Ε, θα πρέπει να κάνουμε το πάντα δυνατό ώστε να αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων εγκλημάτων. Θα πρέπει να επιμείνουμε στην αλήθεια και να καταδικάσουμε οποιαδήποτε πολιτική που μοιράζει, διαχωρίζει, αποκλείει. Χωρίς την αλήθεια δεν ε, υπάρχει ούτε συμβασμός ούτε κερδοσκοπία. Θα πρέπει λοιπόν σε ενθύμηση της Ρεμπρένιτσα ε, φέρω αυτό το λουλούδι προκειμένου να θυμηθούμε πόσο επικίνδυνος είναι ο ακραίος εθνικισμός ε, που χάραξε μια από τις σκοτεινότερες, οφερότερες στιγμές ευρωπαϊκής ιστορίας. Αυτό το λουλούδι ας είναι πραγματικά το σύμβολο μιας Πραγματική πίστη στο μέλλον τη Βοσνίας Ερζεγοβίνη. Κανένα δεν θα πρέπει να χάνει τη ζωή του μόνο επειδή είναι διαφορετικό, επειδή ανήκει σε διαφορετική εθνότητα ή έχει διαφορετική θρησκεία. Θα πρέπει λοιπόν να καταδικάσουμε την ε, τραγωδία τη Ρεμπρένιτσα, τη γενοκτονία τη Ρεμπρένιτσα τον Ιούλιο ε, του 1995 και θα ήθελα όλοι να το κάνουμε αυτό από κοινό Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει κυρία Μπίλντερ. Παρακαλώ από την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία. Έχετε το λόγο. Ε, πρόεδρε, η Σρεμπρένιτσα είναι το πιο τραγικό επεισόδιο της, του πολέμου στη Βοσνία. Ποινικά ε, ήταν βαριέ οι ποινέ που επιβλήθηκαν. Ε, από διεθνή σκοπιά, όλε οι ευθύνε δεν φαίνεται να έχουν ξεκαθαριστεί πλήρω. Και τέλο, πολιτικά. Είναι γνωστό ότι η Σερβία, που βεβαίω δεν εμπλέκεται τα πολύ βαριές οι Σε διεθνές επίπεδο όλοι 2004 εξέφρασε τη λύπη του για μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες. Ε, ο Λαξάνδρ Βούτσις δυστυχώς, τότε πρωθυπουργός της Σερβίας, έγινε δεκτός που ε, είναι λαός και ε, ε, έχει ζήσει στο πετσί του την έννοια γενοκτονία. Η μνήμη της Τρεμπρένιτσα σήμερα θα πρέπει να είναι μνήμη των οικογενειών και όλο αυτό που ε, θυμούνται έναν εκλειπώντα συγγενή, φίλο, σύζυγο, πατέρα που μπορεί να μην γνώρισαν ποτέ. Ε, θα πρέπει επίσης να σκεφτόμαστε όλους αυτούς που διολοφονήθηκαν, τους άνδρες και τις γυναίκες που θρηνούν ε, πέρα από εθνικές διαχωριστικές γραμμές ή κομματικές διαχωριστικές ε, γραμμές. Ευχαριστώ κυρία Μπίλτ. Επόμενος ομιλητές από την ομάδα των Πρασίνων, ο κύριος Ρωμαίο Φραντς. Κυρία Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, στις 11 Ιουλίου του 1995 πριν από 25 χρόνια κατέλαβαν οι Σερβοβόσνοι ε, της Εμπρένισαν και ε, σφαγίασαν πάνω από 8.000 ε, άνδρες και νέους Βοσνίους. Ε, στην καρδιά της Ευρώπης, ε, ε, κάτω από τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας και θα πρέπει να αναρωτηθούμε μα πώς έγινε δυνατό κάτι τέτοιο. Αυτή η αποτυχία βαραίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως η μεγαλύτερη πολιτική της αποτυχία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό με αφορμή αυτή την επέτειο πρέπει να σκεφτούμε γεμάτη ντροπή και πένθος τα θύματα για να μην επαναληφθεί ποτέ κάτι τέτοιο σαν τη Σερμπρέντσα θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Γιατί 25 χρόνια μετά τις συμφωνίες συνευτικές του Ντέιτον, ακόμα και σήμερα ο μίσος, το μίσος και ο εθνικισμός ε, είναι ε, ε, μεγάλα δηλητήρια που κινδυνεύουν να δηλητηριάσουν και, και την κοινωνία και αλλού στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταδικάσει απερίφραστα ε, περιοχές ε, εθνικώς ε, καθαρές. Είναι, ήταν καθαρός ρασισμός αυτό. Δεν είναι εφεύρεση ούτε βοσνιακή ούτε σερβική δεν θα πρέπει τα εγκλήματα πολέμου εις βάρος ανδρών, ε, γυναικών και παιδιών να αποσιωπούνται. Είναι βαριά και βαθιά τα τραύματα. Ε, θα πρέπει να διώκονται ε, φαινόμενα όπως είναι η άνηση της γενοκτονίας και τα εγκλήματα πολέμου. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να έχουμε μια κοινή κουλτούρα μνήμης. Ακόμα είναι τα στερεότυπα πολύ διαφορετικά και ο τρόπος που διδάσκεται η ιστορία είναι διαφορετικός. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ε, τους πολέμους ε, για να υπάρχει συμφιλίωση ε, για αλλαγή. Ιδιαίτερα σε πολλούς νέους η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει χάσει καθόλου την ακτινοβολία της. Γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε τη Βοσνία Ζεγοβίνη προς την ενταξιακή της πορεία και να ενισχύσουμε και τις δημοκρατικές δυνάμεις. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, εκ μέρους του ECR, ο κ. Σέπινγκ το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, σήμερα θυμόμαστε το δράμα της ε, Σεμπρένισσα πριν από 25 χρόνια. Το τραύμα και ε, η πληγή παραμένει ανοιχτή στην Ολλανδία. Είναι η μεγαλύτερη μαζική σφαγή στην Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, τότε ήταν Ολλανδοί, το Ολλανδικό τάγμα, το Dutch Bat που ε, ε, έπρεπε να φυλάξει την πόλη, αλλά ήταν αδύνατη αποστολή. Η εντολή του ΟΗΕ ήταν περιοριστική και ο πλισμός ε, πάρα πολύ ελαφρύς. Εκεί δεν απέτυχε το Dutch Bat, το Ολλανδικό τάγμα, αλλά η διεθνής Ολλανδική πολιτική. Τότε ήμουν εγώ πολιτικός δημοσιογράφος στην Ολλανδία και είχα πει ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι στην πρώην Ιουκοσλαβία. Το ήθελε και η κυβέρνηση και η Βουλή και ο τύπος το υποστήριζε. Οι καλές προθέσεις ε, κατέληξαν σε μια πολιτική ε, απόφαση που στρατιωτικά ήταν ανεφάρμοστη και ε, το τάγμα αυτό ήταν θύμα και όμοιρος των καταστάσεων. Μετά από 7 χρόνια βγήκε η έκθεση που πρέπει να βγάλουμε διδάγματα κι εμείς από αυτή και τιμούμε και τους βετεράνους μας. Μικρή παρηγοριά είναι ότι ο στρατηγός Μλάντιτς ε, τώρα εκτεί ποινή ισόβια κάρτεξη σε μια Ολλανδική ε, φυλακή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον Επίτροπο Βερχέλη, θα πρέπει να αρχίσουμε τον πρώτο γύρο ψηφοφοριών Από τις 9.45 μέχρι τις 11 θα λάβει χώρα η ψηφοφορία με την ίδια μέθοδο ψηφοφορίας όπως εχθές, ονομαστική ψηφοφορία και τα μέλη θα μπορούν να επαληθεύσουν τις ψήφους τους και τα αποτελέσματα ψηφοφορίας συμβουλευόμενοι το έγγραφο που θα δημοσιευθεί, θα αναρτηθεί στο σελίδα του Κοινοβουλίου. Επεξηγήσεις ψήφου θα μπορούν να υποβληθούν γραπτός εξαιρετικά μόνο επεξηγήσει ψήφου που θα πρέπει να περιέχουν το πολύ 400 λέξει. Μόνο αυτέ θα γίνουν αποδεκτέ. Οπότε αρχίζει η ψηφοφορία. Έχετε μέχρι τι 11 να ψηφίσετε. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στι 1 ε, και 30 το μεσημέρι, 13 και 30. Και τώρα το λόγο έχει ο Επίτροπο Βέρχελη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ πολύ που πήρατε αυτό το χρόνο για να συσκεφτούμε και να θυμηθούμε τη γενοκτονία της Εμπρενίτσα. Πρέπει να τιμήσουμε τα θύματα και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς τα θύματα, τις οικογένειες των θυμάτων, όλων εκείνων που έχουν πληγεί από αυτή την απώλεια. Το έγκλημα της γενοκτονίας της Εμπρενίτσα πρέπει να μας υπενθυμίζει συνεχώς ότι αυτές οι πράξεις δεν θα πρέπει ποτέ να επαναληφθούν. Πρέπει να θυμόμαστε επίσης ότι η γενοκτονία δεν συνέβη μόνο στη Σρεμπενίτσα και δεν υπάρχουν διαφορές της γενοκτονίας. Η γενοκτονία είναι γενοκτονία. Ξεκινάμε με το να θυμόμαστε το γεγονός και μετά ακολουθούμε με απότηση φόρου τιμής προς τα θύματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε πίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας ε, διάταξης αφορά την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης. Για αυτή τη συζήτηση δεν έχουμε διαδικασία catch the eye, ούτε μπλε κάρτες γίνονται δεκτές. Έχουμε ένα διάλειμμα, ένα-δύο λεπτά μικρό διάλειμμα, ούτω ώστε να απολυμανθεί το έδρανο του Επιτρόπου και μετά θα δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σχινά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω που ασχολείστε με αυτό το σημαντικό θέμα και ήδη χαίρομαι για την συζήτηση που θα έχουμε. Ο πολιτισμός είναι τμήμα του γονιδιώματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το, η πλούσια η πολιτιστική σκηνή και σκηνή της δημιουργίας ε, είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη και θα πρέπει πάση θυσία να διαφυλαχθεί. Όλοι γνωρίζουμε πόσο ο κλάδος αυτός ε, του πολιτισμού ε, έχει πληγεί. Ο τομέας του πολιτισμού και της δημιουργίας πλήγησαν με πρωτοφανή τρόπο από την πανδημία. 95% του κλάδου αυτού απαρτίζεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από ανεξάρτητους και ελεύθερους επαγγελματίες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι και πολύ συχνά εργάζονται σε πολύ επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε τακτική ανταλλαγή απόψε με τα κράτη-μέλη, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκπροσώπους του κλάδου τους τελευταίους μήνες. Και αυτό για να προτείνουμε κάποιες λύσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε η έκτακτη λύση η λύση εκτάκτου ανάγκη. Μία από τις πρώτες ενέργειες που υιοθετήσαμε είναι να κινητοποιήσουμε κονδύλια του Ταμείου Συνοχής για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που προέκυψαν από την αντιμετώπιση της πανδημίας και τις σχετικές επενδύσεις. Το πακέτο αυτό πρόσφερε ρευστότητα στα κράτη-μέλη και ιδιαίτερη και άνευ προηγουμένου ευελιξία για να κατανείμουν ε, χρηματοοικονομικούς πόρους σε κλάδους που το χρειάζονταν περισσότερο, συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού και της, ε, των τομέων της δημιουργίας. Δεύτερον, άλλη σημαντική έκτακτη πρωτοβουλία είναι το νέο ε, εργαλείο, το πρόγραμμα SURE, για με 100 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του μειωμένου ωραρίου εργασίας ή της ε, μερικής απασχόλησης, για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των εργαζομένων που επλήγησαν από την πανδημία. Και τα κράτη-μέλη θα αξιοποιήσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο το εργαλείο αυτό και τα κονδύλια για να ανακουφίσουν ε, τις ανάγκες των δημιουργών και καλλιτεχνών. Και τρίτον, ε, θεσπίσαμε και το προσωπικό προσωρινό πλαίσιο για τι κρατικέ ενισχύσει, για τη στήριξη τη οικονομία εν μέσω της πανδημίας. Και ο πολιτισμό συμπεριλήφθηκε ω ε, ε, κλάδο που επλήγει ιδιαίτερα από την κρίση μαζί με τον τουρισμό, τις μεταφορέ, ε, τη φιλοξενία και το λιανεμπόριο. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν αυτό το μηχανισμό για τον τομέα της δημιουργίας και τους κλάδους του πολιτισμού. Πέραν όμως αυτών των εκτάκτων μέτρων, Έχουμε λάβει και πολλές ε, επιτούτου δράσεις, ειδικέ δράσεις. Κάποιοι φορείς ε, ε, πολιτιστικών δραστηριοτήτων ανέπτυξαν τις δικές πρωτοβουλίες, πολλά υποσχόμενες για να ξεπεράσουν την κρίση και με το διάλογο αυτό και τις συνέργειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινοβουλίου, κρατών μελών και άλλων φορέων Θέλουμε να εφαρμόσουμε ιδιαικέ πρωτοβουλίε. Για παράδειγμα, ένα από τα καλύτερα παραδείγματα είναι το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Ίδρυμα και το νέο Ταμείο Αλληλεγγύη για τον Πολιτισμό. Μια άλλη πλατφόρμα του κλάδου ήταν η πρωτοβουλία η Ένωση των, των Κλάδων Δημιουργίας. Μια πρωτοβουλία που δημιουργεί ένα κοινό χώρο για όλους τους κλάδους της δημιουργίας και του πολιτισμού και εξασφαλίζει πρόσβαση σε πολλούς πόρου ε, των αντίστοιχων δικτύων. Επίση, πριν από λίγε εβδομάδε. μια διάσκεψη με εκπροσώπους ε, του Συμβουλίου του Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπή και του κλάδου ε, οργανώθηκε σε αυτή την πλατφόρμα. Τώρα έχουμε και ένα εμβληματικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα «Η Δημιουργική Ευρώπη» και εκεί θα ισχύσει μέγιστη δυνατή ευελιξία και ελαστικότητα στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για όλε τι τρέχουσε και μελλοντικέ δράσει. Και μάλιστα παρατείναμε πολλέ προθεσμίε για να διευκολύνουμε την, οριστικο... την οριστικοποίηση τη υποβολή αιτήσεων υπό αυτούς τους χαλιπού καιρού. Και επίση προγραμματίσαμε ειδικά μέτρα για του κινηματογράφου, για παράδειγμα, με επιπλέον κονδύλιο 5 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή κουπονιών για τους κινηματογράφους που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από το lockdown, τα μέτρα απομόνωσης και εγκλισμού. Επίσης, έχουμε και ένα σύστημα στήριξης για τις ε, διασυνοριακά εργαζομένους στον τομέα του πολιτισμού ε, με τίτλο «Ψηφιακό πολιτισμός». Και με το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη θα έχουμε στοχευμένη δράση για να στηρίξουμε τον κλάδο της μουσικής που επίσης πλήγει δυσανάλογα από την πανδημία με την πρωτοβουλία για τη μουσική και 5,2 ε, εκατομμύρια θα αφιερώσουμε φέτος στον κλάδο αυτό για να γίνει ο τομέας της μουσικής ε, πιο, πιο ανθεκτικός μετά την κρίση. Θα ενισχύσουμε λοιπόν τον πολιτισμό και με τη διευκόλυνση των εγγύσεων που θα χρησιμοποιηθεί σε ειδικέ καταστάσεις με μεγαλύτερη ευελιξία, με πίστοση για διακοπέ ή κάποιες, κάποιο μεμονωμένα δάνεια με και καλυμμένε εγγύσει. Έρχομαι τώρα στο σχέδιο ανάκαμψη και στο σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση Επόμενη Γενιά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα είναι πραγματικά συμβολικό και θα ανοίξει το μονοπάτι ε, προς τη συμφωνία για το πολυπόθητο αυτό πακέτο το σχεδίο ανάκαμψης και εκεί θα υπάρχουν ε, ενισχύσεις όχι μόνο για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη αλλά και για άλλα προγράμματα όπως το REACT-EU, τη νέα πολιτική συνοχή, το InvestEU, το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη μεταξύ άλλων. Οπότε πιστεύω ότι θα ήταν λάθος να να θεωρούμε ότι η Δημιουργική Ευρώπη, το πρόγραμμα αυτό είναι το μόνο μονοπάτι για την ανάκαμψη του κλάδου το, στο μέλλον. Έχουμε ένα ευρύ οπλοστάσιο εργαλείων ε, που θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά. Πέραν όμως του, του σχεδίου ανάκαμψης, της δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι έχουμε πολλές δυνατότητες ε, από διάφορες περιπτώσεις όπως το ορίζον Ευρώπη και εκεί υπάρχει ένα κεφάλαιο για το πολιτισμό, την δημιουργία και την κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και εκεί προσφέρονται πολλές ευκαιρίες, μοναδικές ευκαιρίες για τους κλάδους αυτούς και ας μην ξεχνούμε και την κοινότητα γνώσης και καινοτομίας ΚΙΚ, που για πρώτη φορά θα αφιερώνεται και στις, στους κλάδους πολιτισμού και δημιουργίας ε, μέσω του Ινστιτούτου για την Τεχνολογία που εδρεύει στη Βουδαπέστη, κυρία Πρόεδρε. Όλα αυτά λοιπόν τα εργαλεία και οι μηχανισμοί θα συμβάλλουν στην ενίσχυση μιας ισχυρής νέας αρχής του κλάδου αυτού μετά τη δύσκολη εποχή της πανδημίας. Και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και τον τουρισμό. Θα θυμάστε ότι πριν από λίγες εβδομάδες, πριν από ένα μήνα για την ακρίβεια, ε, δημοσιεύσαμε ένα περιεκτικό πακέτο για τον τουρισμό και τα ταξίδια. Ο τομέας του τουρισμού αντιπροσωπεύει το 40%, ε, ο πολιτιστικό τουρισμό είναι το 40% του συνολικού τουρισμού. Και στι αρχέ του καλοκαιριού ε, που ξεκινά και η τουριστική περίοδο, δεν θα ξεχάσουμε και το σημαντικό κεφάλαιο του πολιτιστικού πολιτισμικού ε, τουρισμού. Αυτούς τους δύσκολους καιρούς λοιπόν κυρία Πρόεδρε και κύριε Ευρωβουλευτέ ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, έχει γίνει είδος πρώτης ανάγκης. Ο πολιτισμός είναι τμήμα της κληρονομιάς μας. Ο πολιτισμός, η κουλτούρα είναι ο ε, ευρωπαϊκός τρόπος ζωής και για να τον διαφυλάξουμε, να τον προασπίσουμε και να τον προωθήσουμε θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να συνεργαστούμε για να είναι το νέο αυτό μέλλον του κλάδου όσο πιο λαμπρό γίνεται. Και υπολογίζω στη δική σας βοήθεια, ώστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε, να βοηθούμε, να συνδράμουμε τις δυναμικές κοινότητες των καλλιτεχνών και των δημιουργών μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα διεξαχθεί συζήτηση. Πρώτα η κυρία Σόιντροβα, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ που μπορούμε να δώσουμε αυτή τη μάχη για τον πολιτισμό και τον πολιτιστικό τομέα μαζί. Αυτό δείχνει ότι είναι λογικό να δοθεί αυτή η μάχη. Ευχαριστώ τον κύριο Σχοινά που ανέφερε πολλές δραστηριότητες που συμπληρώνουν τις ήδη γνωστές. Γνωρίζω την Creative Europe, το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, έχει οικονομική σημασία πολιτισμός. 3 με 4% του ΑΕΠ αντιπροσωπεύει στην Ευρώπη. Μη συμπεραβάνοντας το τι έσοδα δίνει στον τουρισμό. Κύριε Σχοινά, το αναφέρατε αυτό στα συμπεράσματά σας. Όλα τα πολιτιστικά μνημεία, οι τοποθεσίες, ε, τα φεστιβάλ, όλα αυτά είναι τουριστικοί προορισμοί. Χωρίς πολιτιστικές δραστηριότητε δεν θα υπάρξει τουρισμός που είναι κινητήρια δύναμη της οικονομίας ε, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό θέλουμε το Creative Europe και το νέο Ταμείο Ανάκαμψης να είναι ανοιχτά ε, εργαλεία, να είναι ανοιχτά και να συμπεριλαμβάνουν αυτές τις δραστηριότητε. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα και εξαρτάται από τα κράτη-μέλη το πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο, τις πλήρες δυνατότητες του για ανάκαμψη και ε, ενεργό χρήση των διαφόρων πολιτιστικών μνημείων, συμπεριλαμβανομένων και των εξάρτητων μέσων ενημέρωσης, της ε, βιομηχανίας των ταινιών. Και κατά κάποιο τρόπο αντισταθμίσουμε τον αντίκτυπο του κορονοϊού από αυτές τις δραστηριότητε, διότι οι συνέπειες του κορονοϊού είναι καταστρεφικές και το ξέρουμε. Εάν δεν ενισχυθεί το Creative Europe, κάτι που ε, επιθυμούμε, θα θέλαμε, κύριε Σχοινά, να το υποστηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να διαθέτει πόρους για τον πολιτισμό, για τι πολιτιστικέ δραστηριότητε και να οδηγήσει επενδύσεις. Το 2018 είχαμε επιτυχή χρονιά πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα θέλαμε να επαναληφθεί εν κατακλείδη. Έχουμε το ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, που είναι ένας ναός για τους χριστιανούς και για τους μουσουλμάνους και τώρα κινδυνεύει. Θα πρέπει μαζί να εξασφαλίσουμε ότι αυτός ο ναός θα παραμείνει μνημείο και θα θυμίζει ότι αυτές οι δύο θρησκείες μπορούν να συμβιώνουν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είναι σημαντικό να περιορίζεστε στο χρόνο αγόρευσης, γιατί αφαιρείται χρόνο αγόρευσης από άλλους. Η κυρία Κάμερβερτ έχει το λόγο εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ωραίε εικόνε είδαμε τη νύχτα τη 22η προ 23η Ιουνίου σε πολλέ γερμανικέ πόλει. Πάνω από 8.000 κτίρια, κέντρα εκδηλώσεων και θέατρα φωταγωγήθηκαν κόκκινα. Βέβαια, αυτή η νύχτα του φωτό έγινε για λιγότερο ωραίου λόγου. Σε πολύ λίγο χρόνο η κρίση του κορονοϊού γκρέμισε όλο τον πολιτισμό και τι εκδηλώσει. Γι' αυτό ενδεχομένω να, έπρεπε να είχε χτυπήσει κόκκινο συναγερμό και στο κτίριο Μπερλεμό. Γιατί φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην έχει καταλάβει απολύτω τα σημεία των καιρών. Και αυτά που μα είπατε, κύριε Επίτροπε, ε, είναι σταγόνα στον ωκεανό ουσιαστικά. Ούτε στο Ταμείο Ανάκαμψη, ούτε στο επόμενο PDP τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πολιτισμό και η δημιουργικότητα λαμβάνονται υπόψη πραγματικά. Ωραία λόγια ζεστά ακούμε, αλλά από ε, λεφτά λίγα και μάλιστα θέλουν να κάνουν και περικοπές από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ ζητώ τουλάχιστον 2% του Ταμείου Ανάκαψης ε, ως διάσωση για τον πολιτισμό και μάλιστα αυτό να καταγραφεί ε, και ε, να είναι υποχρέωση για τα κράτη-μέλη και για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, Creative Europe. Δεν θα πρέπει να ενδώσουμε ως Κοινοβούλιο, να εξακολουθούμε να ζητούμε διπλασιασμό της πρικοδότησης. Ας μην διορθώσουμε μόνο τις ζημιέ που έγιναν προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και καινούργια τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια έχει το λόγο από την ομάδα Renew η κυρία Φάρεγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, κατά τη διάρκεια του lockdown οι καλλιτέχνες ε, και οι δημιουργοί ήταν παρόντες. Μας έδωσαν όνειρο, ε, φυγή, χαμόγελο και δωρεάν, ακόμα και όταν εμείς ήμασταν αποκαρδιωμένοι. Εμείς είμαστε εκεί για αυτούς. Ε, είναι επίγουσα η κατάσταση για τον πολιτισμό, από τη μια μέρα στην άλλη σταμάτησε. Κινηματογράφοι, φεστιβάλ, μουσεία, θέατρα, μνημεία είναι τα πρώτα που έκλεισαν και τα τελευταία που θα ανοίξουν μετά από πολλούς μήνες απολειών και αβεβαιότητας, την οποία δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως ανακοινώνοντας τα γελία ποσά που δίνονται ε, στα νέα προγράμματα για τη δημιουργική Ευρώπη. Μόλις είναι 8% το Κοινοβούλιο ζητούσε διπλασιασμό. Ας ε, θυμηθούμε ότι μόνο 0,14% αφιερώνει η Ευρώπη στον προϋπολογισμό της για τον πολιτισμό. Μα ε, ε, είναι ανησυχητικά αυτά τα σημάδια. Θα πρέπει η ανάκαμψη του πολιτισμού να περάσει από την Ευρώπη. Θα πρέπει να κινητοποιήσετε όλους τους μηχανισμούς και το πρόγραμμα SURE ε, για ε, όσους είναι σε αναστολή λειτουργίας και το Next Generation EU για να χρησιμοποιηθεί ε, για την ενίσχυση του κλάδου που έχουν επιχειρήσεις εκεί διαφόρων μεγεθών αυτοπασχολούμενους 4% του επ. Μετά την επίγουσα κατάσταση θα πρέπει η Ευρώπη να είναι φιλόδοξη και να δείξει ότι είναι αναντικατάστατος ο πολιτισμός, ποια είναι η πολυμορφία μας και πόσο μας ενδιαφέρει η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός. και η πολιτιστική κληρονομία και μπορούμε ε, ε, ε ευκαιρίες να του δώσουμε και μεγάλε ευρωπαϊκέ συμπαραγωγέ. Ε, ε, ε, και στο, στην Πράσινη Συμφωνία έχει χώρο για τον πολιτισμό. Τέλο, κύριε Επίτροπε, α έχουμε αυτή τη φιλοδοξία για να ενισχύσουμε την Ευρώπη και να δώσουμε μια πηξίδα στι ευρωπαϊκέ αξίε. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη διάσκεψη για την Ευρώπη και ο πολιτισμό, στο διάλογο με του πολίτε. Αλλά πρώτα απ' όλα και για να είναι ο πολιτισμό το μέλλον τη Ευρώπη, θα πρέπει η Ευρώπη να δώσει μέλλον στον πολιτισμό. Σας ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Αντώνιο Νταρέκ, μέρο ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα του ID, κυρίω και το κίνημα για το Σαβίνι, ε, θέλουμε να εμποδίσουμε την καταστροφή. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε εμεί την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τη βελτιώσουμε, γιατί γι' αυτό μα κατηγορούσαν. Στι 26 Οκτωβρίου του 2019, εγώ έστειλα μία επιστολή στον πρόεδρο, τον κύριο Σασόλη, ζητώντα να ξεκινήσει η συνταγματική ενθεώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση που έλαβα από τον πρόεδρο ε, δήλωσε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν αυτή την κατεύθυνση υπογραμμίζοντας τον κεντρικό χαρακτήρα που έχει ο πολιτισμός στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να, ε, θα πρέπει να ξαναγεννηθεί. Δεν θα πρέπει να είναι η Ευρώπη των εθνών, αλλά η Ευρώπη των λαών. Να υπενθυμίσουμε το, το λαό της Βενετίας και του Φρίουλη, ε, της Καταλωνίας, τους Βάσκους, τους Βρετόνους κλπ. Δεν θα πρέπει να μιλάμε για ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά ένα άθροισμα πολιτισμού λαών που απαρτίζουν την Ευρώπη. Η προσπάθεια να αφημώσουμε τις, τις διάφορες ιδιαιτερότητες δεν μπορεί να οδηγήσει σαν απόφευκτη χρεοκοπία του, του εγχειρήματο του ευρωπαϊκού, κάτι που δεν θέλουμε. Σεβόμαστε πλήρω τον πολιτισμό, την ιστορία των διαφόρων χωρών. Μόνο μέσα αυτού του σεβασμού θα πετύχουν πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό πολιτισμό μπορεί να δημιουργηθεί πέρα από τα εθνικά συμφέροντα που δημιουργούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ταυτότητε οδηγούν σε προστιθέμενη αξία που μεγαλώνουν και κάνουν την Ευρώπη ε, μοναδική με 500 εκατομμύρια πολίτες θα πρέπει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός να αποτελέσει προτεραιότητα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών και να είναι βασική αρχή, ε, συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρξει Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς το σεβασμό των διαφόρων κανόνων, των διαφόρων ταυτοτήτων, χωρίς το σεβασμό της Λαϊκή Βούληση, αν, αν τελικά ίσω πηγιστρέφεται καμιά φορά κατά τη Ευρωπαϊκή ε, γραφειοκρατίας η βούληση του λαού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε πίτροπε. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τον πολιτισμό. Αυτό είχε πει ο Ζάμονε και έχει μεγάλη σημασία τώρα που αναζητούμε να βρούμε τον τρόπο ζωή που πρέπει να ακολουθήσουμε στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια τη κρίση του COVID, ο πολιτισμό ήταν παντού, σε όλα τα σπίτια. Στον περιορισμό ε, μα ανακούφισε ε, ο πολιτισμό. Ήταν ένα στοιχείο ζωτική σημασία για μια κοινωνία. Ο πολιτισμό εκφράζει και εκπροσωπεί και σε κάνει να κάνει την υπέρβαση και συνδέει τις γενιές, τους ανθρώπους, τις γλώσσες, διασκεδάζει, κεντρίζει τη φαντασία, τα μουσεία, τα θέατρα, αίθουσες χορού, ε, βιβλιοθήκες, μας ενώνει ο πολιτισμός και μπορούμε να καταλάβουμε ένα στον άλλο μέσω του πολιτισμού και να ε, καταργούμε τις διακρίσεις και ενισχύουμε την αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη, τη δημοκρατία, την ισότητα και την αλληλεγγύη που είναι ιδρυτικές αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ακόμα βλέπουμε ότι είναι δήλωση αγάπη που κάνω εγώ προ πολιτισμό και προ εκείνου και εκείνε που την κάνουν να ζει. Η κρίση, έλλειψη αναλογική και φιλόδοξη αντίδραση των πολιτικών μα έπληξε πολύ σκληρά σε αυτού του ανθρώπου που παράγουν πολιτισμό και είναι το επάγγελμά του. Είναι τεχνικοί, δημιουργοί, ε, συγγραφεί, καλλιτέχνε. Για όλου αυτού η ανάκαμψη θα πρέπει να είναι η στιγμή που δεν θα πρέπει να είναι παράπλευρη ε, δραστηριότητα πολιτισμός, θα πρέπει να έχει προτεραιότητα πολιτισμός σε επίπεδο πολιτικό και χρηματοδοτικό. Θα πρέπει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα να μπει στο επίκεντρο πολιτισμός. Είναι, θέλουμε λοιπόν να αφήσουμε πίσω έναν κόσμο με κρίση και πολέμους για τα παιδιά μας. Λοιπόν, όπως είπε και ο Λιβιέ πει, θα πρέπει να αρπάξουμε τώρα αυτή την ευκαιρία που μα προσφέρεται, αυτή να ξαναδημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα εντό του οποίου ο πολιτισμό δεν θα είναι πολυτέλεια, αλλά ένα καθήκον. Επιτακτικό. Λοιπόν, οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητή, ο κύριος Τζαμπάσκη, εκ μέρου του ECR. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, Αναμφίβολα η συζήτηση αυτή είναι πολύ σημαντική και το θέμα είναι μείζονος σημασία. γιατί ο πολιτισμός ε, βρίσκεται στη ρίζα της ταυτότητάς μας και του αυτοπροσδιορισμού μας. Γι' αυτό και τέτοιους καιρούς θα ήθελα να έχουμε μια σοβαρή συζήτηση για το τι θα πρέπει να θαρρύνει και να προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ακολουθήσουμε τον ολιστηρό πάλι δρόμο και θα ενθαρρύνουμε υπερεθρικά πολιτιστικά τικός μαρξιστικά σχέδια που θα επιχειρήσουν ε, να προστατεύσουν το ευρωπαϊκό μόρφωμα χωρίς ε, εθνική ταυτότητα, χωρίς ε, ε ουσιαστικές καταβολές πολύ αμφιβάλλω ότι ένα τέτοιο υπερεθνικό μόρφωμα θα τα καταφέρει. Γιατί εμείς οι Ευρωπαίοι ε, είμαστε σήμερα αυτό που είμαστε, γιατί έχουμε την παράδοση που μας χαρακτήρισε για αιώνες, τη χριστιανοσύνη, διάφορα είδη χριστιανοσύνης και όταν μιλούμε για τις καταβολές μας, για τις ρίζες και την προέλευσή μας, δεν μπορούμε να ξεχνούμε την Αγία Σοφιά και την Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι τυχαίο που ε, αναφέρεται ως η μητέρα όλων των εκκλησιών. Και δεν μπορεί η Τουρκία να ε, θεωρεί την Αγία Σοφιά εσωτερικό εθνικό ζήτημα, εγχώριο. Είναι κοινό στοιχείο της δικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς. Παρακαλώ να το επισημάνετε στον πρόεδρο Ερτογκάν. Δεν μπορεί να αποδοπατά τα ευρωπαϊκά έθνη ο κύριος Ερτογκάν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρου ε, τη ΓΚΟΕ, Ανατολική Αριστερά, το λόγο έχει ο κύριο Κιζίλ Γιουρέκ. μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξασφαλίζεται μόνο με την κοινή αγορά. Ούτε μπορεί να χτιστεί το αίσθημα του εμεί ή του μαζί μόνο με το κέρδο. Αν έχει κάτι που φέρνει μαζί του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι η κουλτούρα και ο πολιτισμό. Δυστυχώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει τη δέουσα σημασία στον τομέα τη κουλτούρα είναι γεγονό ότι το τομέα τη κουλτούρα μπήκε βάναυσα κατά τη διάρκεια τη πανδημία του κορονοϊού. πολλά κράτη μέλη όπω και η χώρα μου η κύπρος ουσιαστικά έχουν ξεχαστεί τον τομέα του πολιτισμού και του ανθρώπου του οι οποίοι ανάμεναν εδώ και μήνε κάποια στήριξη αρκούνται όμω σε υποσχέσει. Ζητούμε σημαντική ενίσχυση του χρηματοδοτικού προγράμματο για τον πολιτισμό την περίοδο 2021-2027 και ενό επαρκού χρηματοδοτικού πακέτου κίνητρων για πολιτιστικούς δημιουργούς σε όλη την ευρώπη. ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα στηρίξει τις ομάδες πολιτιστικής δημιουργίας. μόνο έτσι μπορούμε να επενδύσουμε στο αίσθημα του εμείς και στις γενιές του μέλλοντος. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Μιγιάν μόνο εκ μέρου του ΕΛΚ. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το Ταμείο Ανάκαμψη και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα, δεν θα πρέπει να ξεχνούν την πολιτιστική διάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Erasmus Plus και η Δημιουργική Ευρώπη θα πρέπει να έχουν αυξημένα κονδύλια. Όλοι αυτό ζητούμε και σε αυτό προσβλέπουμε. Επίση, θα πρέπει να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά, που όπω είπατε, κύριε Αντιπρόεδρε, δραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να προσελκύσει τον τουρισμό, ένα τομέα που έχει πληγεί τα μάλα από την πανδημία. Το πρόγραμμα της Συμβουλίου της Ευρώπης για, ε, για τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά μονοπάτια είναι σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θα πρέπει να συμβάλλουμε στη χρηματοδότησή του. Και του χρόνου το πρώτο αυτό μονοπάτι, ο δρόμος του Σαντιάγο, θα εορτάσει το ιερό ε, έτος, επαιτειακό έτος. Επίσης, ε, το 2021 θα έχουμε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις τις σημαντικότερες στην Ευρώπη και θα πρέπει να βοηθήσουμε και από τη δική μας πλευρά. Οι δρόμοι του Σαντιάγο είναι δρόμοι της Ευρώπης, ε, περνάνε όλες τις χώρες της Υπήρου και για αιώνες ολόκληρους πολλοί, πολλοί πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφταναν στο Σαντιάγο Κομποστέλα, συμβάλλοντος στη δημιουργία και στην εξάπλωση μιας ευρωπαϊκής κουλτούρας αλλά και μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Και επίσης ε, θα ήθελα να προσυπογράψω και εγώ την ερώτηση της κυρίας Σόιντροβα δεν θα πρέπει να αντιταχθούμε σε αυτό το σχέδιο να χαρακτηριστεί τζαμία για Σοφιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Βίκτορ Νεγκρέσκου, εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Είναι πολύ σημαντική, αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση αυτή για τον τομέα του πολιτισμού και τη δημιουργία στην Ευρώπη που επλήγει από την πανδημία του COVID. Ε, χιλιάδες άνθρωποι που απασχολούνται στον τομέα αυτό δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν στις αλλαγέ που επέφερε η πανδημία και οι εθνικές ε, λύσεις δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων για να προστατεύσουν αυτούς τους κλάδους της δημιουργίας και του πολιτισμού. Κάναμε πολλές προσπάθειες για να πείσουμε τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν και δυστυχώς μέχρι στιγμής ε, οι καλλιτέχνες μας είναι ξεχασμένοι της πανδημίας. Το ίδιο συνέβη και στη Ρουμανία. Τίποτα δεν κάναμε για τις 3.500 εργαζομένους στον κλάδο αυτό που συμβάλλουν στη δημιουργία του 10% του ΑΕΠ. Θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαφή μέτρα για την υποστηρίξη του κλάδου. Θέλουμε 2% του σχεδίου ανάκαμψης να αφιερωθεί στον τομέα της δημιουργίας και του πολιτισμού. Αντίστοιχε δράσει θα πρέπει να αναλάβουν και τα κράτη-μέλη. Και το ψήφισμά μα είναι η τελευταία έκκληση για την διάσωση του κλάδου. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην κοφεύσει στι χιλιάδε φωνέ των εργαζομένων που απασχολούνται στον κλάδο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενο συνάδελφο. Λυπάμαι, λυπάμαι. Δεν υπάρχει η διαδικασία της γαλάζιας κάρτας στην συζήτηση αυτή. Διαδικαστικό. Να παραταθεί συζήτηση, ζητώ. Είναι η πρώτη συζήτηση που διεξάγεται για το θέμα του πολιτισμού και δίνεται 30 λεπτά, που είναι αστείο να γίνεται μια τέτοια συζήτηση και δεν επιτρέπεται η γαλάζια κάρτα και μας σέρνεται σαν να είμαστε κοπάδι δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό, δεν αρκεί για το σημαντικότατο θέμα που συζητάμε. Η ε, Πρόεδρος, ευχαριστώ για αυτό που λέτε, για την άποψή σας. Γι' αυτό προσπαθώ να σας παρακαλέσω να σεβόσαστε το χρόνο αγόρευσή σας. Λόγω ε, των περιορισμών της διερμηνίας δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Ελπίζουμε να επανέλθουμε στην κανονική λειτουργία μας σύντομα και να έχουμε πιο μακροσκελή συζητήσεις. Ο κύριος Νίνας έχει το λόγο εκ μέρους των ε, Πρασίνων. Παρακαλώ αν έχει την καλοσύνη να σεβαστείτε το χρόνο αγόρευσή σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχετικά περιορισμένη στις δυνατότητες και τις εξουσίες ε, που έχει για ε, τον πολιτισμό και απευθύνομαι στο Συμβούλιο που λάμπει δια της απουσίας του. Η κυρία Μέρκελ δεν είπε το παραμικρό για ε, τον πολιτισμό εκτός από το γεγονός ότι είναι τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Μπετόβεν. Και ε, να πω ε, κάτι που είπε ο Μπετόβεν. Ο, ο κόσμος που δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει πολιτισμός είναι καταδικασμένος. Όποιος γιορτάζει την κληρονομιά του Μπετόβεν αλλά δεν ε, ενισχύει τον πολιτισμό θα γνώριζε μόνο ε, την περιφρόνηση από τον Μπετόβεν. Δεν έχετε καταλάβει σε ποια ε, κατάσταση βρίσκεται ο πολιτισμός, καταστροφικός. Ενωμένη στην πολυμορφία είναι το σύνθημά μας. Ποια πολυμορφία κινδυνεύει να εξαφανιστεί αν δεν βοηθήσουμε τη δημιουργική βιομηχανία στην Ευρώπη για να σας ε, εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Ε, χωρίς γραφειοκρατία, ελάχιστο εισόδημα για τους καλλιτέχνες, ευρωπαϊκή κοινωνική ε, εγγύηση για τους καλλιτέχνες. Τι, θα γνωρίζετε την περιφρόνηση όλων των καλλιτεχνών, αν τιμάτε μόνο τους νεκρούς καλλιτέχνες και όχι τους ζωντανούς. Ευχαριστώ. Πελτιέ από την Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Επτά εκατομμύρια καλλιτέχνες, εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες στον ε, πολιτισμό. Ε, ε, αυτοί οι εφευρέτες ψυχής, όπως έλεγε και ο ε, ε, κινδυνεύουν και κρέμονται από τις ανακοινώσεις των κρατών και της Ένωσης. Αναβάλλονται, ματαιώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είναι συχνά ο φτωχός συγγενής και είδαμε πόσο υπέφεραν από το lockdown ε, μέσα σε δύο μήνες το Λούβρο δέχτηκε 10 εκατομμύρια εικονικές επισκέψεις. Ε, ο πολιτισμός δεν είναι πρόθεση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Είναι κοινό αγαθό που χτίζει μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο ανεκτική. Ας επιλέξουμε να απαντήσουμε με το πολιτισμό στις απειλές ε, περιχαράκωσης και ταυτότητας. Μερικοί βουλευτές μόνο για ταυτότητα μιλάνε και ξέρουμε πόσο είναι απειλή να έρθουν οι εθνικιστές στην εξουσία. Ξαναδείτε τον προπολογισμό και αυξήστε το Creative για να βοηθήσουμε τους καλλιτέχνες. Ο Μίλαν Κούντερα έλεγε ότι ο πολιτισμός είναι η μνήμη του λαού. Η συλλογική μας ε, συνείδηση για την ιστορική ε, συνέχιση ενός τρόπου σκέψης και ζωής. Σταματήστε τη λιτότητα και ξανασκεφτείτε την ε, χρηματοδότηση της δημιουργικής δραστηριότητας και παραγωγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπεν Χουμέα, παρακαλώ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, μιλώ για πρώτη φορά στην Ολομέλεια από το Φλεβάρι και θα ήθελα να στείλω τα βαθύτατα συλληπιτήριά μου προς τις οικογένειες των θανόντων από το COVID-19 και να εκφράσω την ικανοποίηση μου και την, ευχαρίστηση, και την ευχαριστία μου σε όσους εργάζονται για την καταπολέμηση της πανδημίας. Μιλούμε για το πολιτισμό, στρατηγικό τομέα, σημαντικό στην Ευρώπη. Ακούσαμε ε, διάφορες ε, τοποθετήσεις και ποσά. Θέλω να μιλήσω εδώ ε, για την πολιτιστική ταυτότητα της Ευρώπης, για τις ε, Ιουδεοχριστιανικές αρχές. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπερασπιστεί αυτή την ευρωπαϊκή ταυτότητα και τις δυτικές αξίες. Και αυτό βλέπουμε τι γίνεται με την Αγία Σοφιά που θέλουν να την κάνουν τζαμί ή ε, με τις επιθέσεις που είδαμε στα μνημεία στην Ευρώπη από ολοκληρωτικά κινήματα που προωθούνται από εκείνους που θέλουν να επιτεθούν στην ταυτότητά μας, στον πολιτισμό μας και στις αξίες μας. Θα πρέπει να το διατρανώσουμε μόνο και να βοηθήσουμε τον πολιτισμό, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε έτσι και τη δημοκρατία και τις ελευθερίες στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος είναι ο κύριος Μερίλιο, εκ μέρους των Σελιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να λησμονηθεί. Οι τομέες δημιουργική και καλλιτεχνική στατική σημασία χρειάζεται ένα νέο deal της στον πολιτιστικό τομέα Από τα ξεκινά από τι κατεπίγουσε ανάγκε που δημιουργήθηκαν σε αυτή την εποχή, την αποστασοποίηση, την κοινωνική, κενά θέατρα και κινηματογράφου. Πολιτισμό σημαίνει περιεχόμενο αλλά και εργασία πολύ συχνά επισφαλή η πρόσφατη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επόμενο πολιτέ ε, δημοσιονομικό σχέδιο δεν ανταποκρίνεται στο ύψο τη πρόκληση. Θα πρέπει να διπλασιαστεί το προπολογισμό για τη Δημιουργική Ευρώπη. Θα εξακολουθεί το ζητά το Κοινοβούλιο. Με το Next Generation μπορούμε να δημιουργήσουμε συνδέσει με άλλου πόρου χρηματοδότηση, να δημιουργηθούν συμπράξει και συνέργειε. Η πολυσχηδή ε, πολιτιστική δραστηριότητα τη Ευρώπη πρέπει να προωθηθεί. Πρέπει να ενισχύσουμε τα προγράμματα που υπάρχουν όπως στη Δημιουργική Ευρώπη και να μεγιστοποιήσουμε τη δυνατότητα του Recovery Fund. Θα πρέπει να βρούμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Χινάς έχει το λόγο. έχει το λόγο κύριε Χινά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι συμφωνούμε απόλυτα όσον αφορά τη διάγνωση της καταστάσεως όσο και τις ε, δράσεις που θα πρέπει να δρομολογηθούν για να ανακοφιστούν οι συνέπειες της ε, πανδημίας σε έναν από τους τομείς που είναι ο πιο δημιουργικός, ο πιο δυναμικός που συνδέεται περισσότερο με τις παραδόσεις μας, με την ε, ποικιλομορφία του πολιτισμού μας. Σημείωσα επίσης τις ανησυχίες σας για τον προϋπολογισμό, για τα προγράμματα. Ξέρετε ότι όσον αφορά τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό, αυτές οι συζητήσεις πάντα, μα πάντα είναι περίπλοκες. Αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι αυτό που βρίσκεται επιτάπητος είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή που θα μπορούσαμε να προτείνουμε υπό τις παρούσες περιστάσεις και επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας την αισιοδοξία μου. Πιστεύω την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια πολύ μεγάλη ιστορική συμφωνία για το πακέτο ανάκαμψης και θα είναι ένας καλύτερος τρόπος για να συμβολήσουμε ε, την επαναφορά της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης και της απασχόλησης. Σημείωσα την παραδοσιακή συζήτηση για το τι αντιπροσωπεύει σήμερα η ευρωπαϊκή κουλτούρα. Είχα και την ευκαιρία στην ακρόασή μου να πω ότι βλέπω ότι είναι πολύ πλούσια η πολιτιστική μας κληρονομιά. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο επειδή υπάρχει το Homo Europaeus, ένας, ένα, ο άνθρωπος που σκέφτεται παρομοίως και επιβάλλει εκείνος ή εκείνη τις αξίες του, τις αξίες της σε όλους τους άλλους. Βλέπω τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σαν ένα καθρέφτη. Ένα καθρέφτη ποικιλομορφίας ένα καθρέφτη που αντικατοπτρίζει τον πλούτο αυτού που εκπροσωπεί η Ευρώπη από πλευρά γλώσσα, ιστορία, παράδοση, πολιτισμού, λογοτεχνία, τεχνών. Και αυτό είναι που κάνει την Ευρώπη μοναδική στο σημερινό αβέβαιο και τολμώ να πω πιο σκοτεινό κόσμο. Κάτι άλλο θα ήθελα να πω επίσης για την Αγία Σοφία. Σημείωσα το ενδιαφέρον σας και το μοιράζομαι. Η Αγία Σοφία είναι ένα σύμβολο. Σύμβολο διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό. Διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου. Αποτελεί ένα τμήμα του πολιτιστικής κληρονομίας UNESCO. Είναι ένα μουσείο, είναι ένα σύμβολο. Σύμβολο μιας πόλης. Που αυτή καθε αυτή η πόλη είναι ένα σύμβολο αυτό που, που θα θέλαμε να δούμε σαν μία από τις αξίες που θα έπρεπε να επικρατούν στον κόσμο. Η Τουρκία είναι ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας του ΙΕ για τη Συμμαχία των Πολιτισμών και ήδη έχει αναλάβει συμβασιακές υποχρεώσεις σε αυτό το πλαίσιο. Είναι παγκόσμιο μνημείο η Αγία Σοφία. Το να διατηρηθεί το καθεστώς του μνημείου αυτού που αναγνωρίζεται και διεθνώς και δημοσίως είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί αυτό το καθεστώς. Διαφορετικά θα αιμονεμηθεί η ανοιχτή τοποθέτηση και η ανοχή που επικρατεί στη Τουρκία. Να επιθυμίσω ότι το 2010 η, η πόλη που φιλοξενεί την Αγία Σοφία ήταν ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα και ο Πρωθυπουργό της Τουρκίας τότε, ο Ρατζίπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε πει «Αυτή είναι μια ευρωπαϊκή πόλη με την καρδιά της, τον πολιτισμό της και τον πολιτισμό της και το λαό της, το παρελθόν της, το μέλλον της, πάντα έβλεπε προς την Ευρώπη αυτή η πόλη. Η Κωνσταντινούπολη διαμόρφωσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και διαμορφώθηκε από αυτόν. Πρωθυπουργό Ερντογάν, έτος 2010. Αυτό είναι το πνεύμα που θέλουμε να επικρατήσει. Αυτό περιμένουμε από τον πρόεδρο Ερντογάν μετά από 10 χρόνια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και με την παρέμβαση του Επιτρόπου Σχοινά ολοκληρώνουμε το θέμα αυτό, τη δήλωση της Επιτροπής για την πολιτιστική ανάκαμψη Ευρώπης. Ευχαριστώ θερμά τον Επίτροπο για την παρουσία του και τη συμμετοχή του στη συζήτηση. Η ψηφοφορία για το θέμα αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο, όπως γνωρίζετε. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Περιμένουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Επίτροπο, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Έλαβε θέση Επίτροπος. Καλημέρα σας και πάλι. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα το ρόλο της πολιτικής συνοχής στην αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του COVID-19. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δεν προβλέπεται για τη συζήτηση αυτή, ούτε διαδικασία κατσδιάη, ούτε υποβολή ερωτήσεων με την μπλε κάρτα. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον συντάκτη της προφορικής ερώτησης, στον συνάδελφο Γιουνούσο Ομαρτζή, για πέντε λεπτά για να μας την παρουσιάσει. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, αγαπητή Ελίζα Φερέα, αγαπητοί συνάδελφοι, το πρόσωπο της Ευρώπης έχει παραμορφωθεί από την κρίση της COVID-19. Όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες πλήττονται σφοδρά. Η ανεργία εκτοξεύεται, οι ε, χρεοκοπίες πληθύνονται, οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν πληγεί σφοδρότατα. Κανένας ε, κλάδος και καμία περιφέρεια δεν έχουν γλιτώσει και οι ε, οικονομικές προβλέψεις είναι μάλλον καταστροφικές. Η κρίση αυτή είναι ε, σκληρή ε, απόδειξη ε, του ευάλωτου χαρακτήρα μας. Σήμερα η ανάκαμψη δεν είναι επιλογή, είναι επιταγή. Περισσότερο από ποτέ τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να κρατήσουν μία αρχή και μία ρότα της συνοχής σε αυτή την ε, υγειονομική καταστροφή που μένετε, ε, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μόνη η ευρωπαϊκή πολιτική που κατάφερε να βοηθήσει όλα τα κράτη-μέλη είναι η πολιτική συνοχής. Η πολιτική αυτή βοήθησε να δημιουργηθούν ε, ε, προβλέψεις ε, για την ενίσχυση εργαζομένων που ήταν σε αναστολή, για να βοηθηθούν τα νοσοκομεία σε εξοπλισμό, ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όπως και η Επιτροπή μας Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, αναλάβαμε τις ευθύνες μας και εγκρίναμε την νομοθεσία με κατεπίγουσα διαδικασία αρχίσαμε και την ομοθετική δουλειά για το React-EU. Εδώ ε, την Τετάρτη ε, στην Ολομέλεια η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Ούρσουλα Φόντα Λάιεν μαζί με όλους τους προέδρους των πολιτικών ομάδων συνηγόρησαν υπέρ της ανάκαμψης που να βασίζεται στη συνοχή. Στο εξή λοιπόν περιμένουμε τα λόγια αυτά να μεταφραστούν σε έργα και να εγγραφούν σε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Περιμένουμε λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποδειχθεί στο ύψος των υποσχέσεων και των προσδοκιών στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής. Κυρία Επίτροπε, στο νέο μέσο Next Generation EU προτείνονται κάποιες χρηματοδοτήσεις. Είναι ένα καλό βήμα πρόοδου προς τη σωστή κατεύθυνση, ακόμα και αν το κύριο βόλιο μα περίμενε πιο γενναία πρικοδότηση. Παρ' όλα αυτά, ε, η πολιτική συνοχής ε, πραγματικά υποφέρει πολύ από τη νέα πρόταση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ε, προβλέπεται μείωση κατά 12% σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η πολιτική συνοχής είναι πρωταγωνιστής σε όλες τις περιφέρειες Ευρώπης είναι μια πολιτική που βασίζεται στην τοπική πραγματικότητα και συμμετέχει στην τοπική οικονομία. Γι' αυτό είναι απόλυτη απαραίτητη η στήριξη κατάλληλη κάθε φορά ε, για να μην υπάρχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες. Περιμένουμε μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη απλούστευση. Και σε αυτούς τους δύο στόχους θα είμαστε στο πλευρό σας για να σας ε, διευκολύνουμε. Από τότε που καταθέσαμε την προφορική μας ερώτηση μέχρι σήμερα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ε, έχουν ε, έρθει πολλές απαντήσεις αλλά παραμένουν πολλά και τα ερωτηματικά. Θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θα επαγρυπνούμε έτσι ώστε τα 350 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης ε, μέσω επιχορηγήσεων ελπίζουμε να καλύψει τους στόχους της συνοχής. Γι' αυτό σας ερωτούμε, κυρία Επίτροπε, τι ρόλο επιφυλάσσεται στην ε, συνοχή εντός της ανάκαμψης και το ευρωπαϊκό εξάμεινο πώς θα προσανατολίσει τα κονδύλια προς τη συνοχή. Δηλαδή η προτεραιότητα να δίνεται στις περιφέρειες, στις λιγότερο ανεπτυγμένες αλλά και σε εκείνες που επλήγησαν πιο σφοδρά από την κρίση. Με ποιο τρόπο επίσης το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα στοχεύσει ακριβώς ε, στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης τις περιφέρειες, ε, τις ομάδες και τους κλάδους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη έτσι ώστε οι νησιωτικές περιφέρειες και οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες να μην εγκαταληφθούν στη μοίρα τους. Και τώρα που όλα τα κράτη-μέλη θα ε, προσφύγουν στο δανεισμό Πώς σκέφτεστε να εξαιρέσετε τις πολιτικές συνοχής το 2021-2027 από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάκαμψης και Ανάπτυξη. Συγγνώμη. Ελπίζουμε να επιτευχθεί μια καλή συμφωνία στο Συμβούλιο. Όλοι μας. Σε περίπτωση που ικανοποιηθεί το Κοινοβούλιο από τη συμφωνία αυτή, η Επιτροπή μας Περιφερειακής Ανάπτυξης και όλοι οι εισηγητές θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας για να ε, ε, προχωρήσουμε ε, σε μια διαπραγμάτευση μέχρι τα τέλη του έτους, έτσι ώστε το 2021 να μην είναι μια χαμένη χρονιά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Μαρτζή. Μας κάνατε μια εισαγωγή σε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση για το ρόλο της πολιτικής συνοχής στην αντιμετώπιση των ε, συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Έχουμε εδώ στη συζήτηση παρούσα την Επίτροπο Ελίζα Φερέιρα, την οποία καλωσορίζω και την ευχαριστώ που ήρθε και ε, μας έδωσε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε και με μεγάλη χαρά σας δίνω το λόγο κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά και τον Πρόεδρο Μαρζή, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση ε, σε αυτή την πολύ επίκαιρη συζήτηση. Μου δώσατε ψήφο εμπιστοσύνη στο παρελθόν και μου αναθέσατε το καθήκον να ε, εργαστώ για μια ισχυρότερη κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή στην Ευρώπη. Και μάλιστα η υποστήριξη των περιφερειών θα μα επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τι ε, σημερινέ και τι μελλοντικέ προκλήσει. Οι σημερινέ προκλήσει είναι ακόμη σημαντικότερε. Ε, Πρόσφατε οικονομικέ προβλέψει Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι οικονομικέ συνέπειε τη κρίση θα είναι περισσότερε από τι αναμενόμενε. Η ανάκαμψη του χρόνου θα είναι χαμηλότερη από την αρχικά προβλεπόμενη. Και η κίνδυνη ύφεση είναι σημαντική. Ε, διαφορές, ασυμμετρία, κατακαιρματισμός ε, είναι απειλές ε, που επικρεμούνται επί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν όλοι από κοινού να βρούμε την πολιτική βούληση και να δείξουμε ηγετικό ρόλο προκειμένου να θέσουμε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει θέσει επιτάπητος ε, ένα πακέτο ανάκαμψης ε, ιδιαίτερα φιλόδοξο και πρωτοφανές ε, περικοδοτημένο που θέτει τη συνοχή και την αλληλεγγύη στο επίκεντρο του. Και σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση αυτής της πρότασης. Οι δύο τα δύο ψηφίσματα που υποστηρίχθηκαν από ευρεία πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν τολμηρέ προτάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια θα πρέπει να τελειοποιήσουμε και να οριστικοποιήσουμε κάποια ζητήματα, αλλά αυτό είναι τμήμα τη δημοκρατική διαδικασία. Το κρισιμότερο, όπως αναφέρατε, και το πιο σημαντικό είναι να μην ε, ολιγορούμε στις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να, καταλήξουμε στη συμφωνία και για τους δύο μηχανισμούς ε, ε, από το και στο πολίτε δημοσιονομικό πλαίσιο 21-27 και στο Next Generation EU με πλήρη σεβασμό της κοινοτική μεθόδου. Έχοντα υπόψη ότι κάθε μέρα που χάνουμε ε, χωρίς να λαμβάνουμε δράση είναι ε, απώλεια μιας ζωής, μιας επιχείρησης, μιας θέση απασχόλησης που χάνεται χωρίς υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που το επισημάνατε κύριε ότι η συνοχή έχει κέρια σημασία για να καταπολεμηθούν οι διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών και οι και για να εξασφαλιστεί ε, ένα πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού που είναι απαραίτητο για μια εύρυθμη εσωτερική αγορά. Θέλουμε τι κατάλληλε επενδύσει για την πράσινη και την ψηφιακή μας ανάκαμψη και δράσαμε άμεσα με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με την υποστήριξη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και προπολογισμού και μάλιστα με τις δύο επενδυτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του COVID κινητοποίησαμε περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια της συνοχής, όπως μας είπατε και εσείς κύριε Μαρζή. Έτσι αγοράσαμε χειρουργικές μάσκες, αναπνευστήρες, ε, σώσαμε θέσεις απασχόλησης και επιχειρήσεις και στηρίξαμε και τα συμπιεσμένα δημόσια οικονομικά. Ήταν έκτακτη ανάγκη. Βέβαια, τώρα χρειαζόμαστε περισσότερε δράσει. Γενικώ, το Ταμείο Ανάκαμψη και η δέσμη μέτρων για τις ανάκαμψη προσφέρει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια που προστίθενται στη συνοχή. Τα μισά θα προέλθουν από το React EU. 55 δισεκατομμύρια ευρώ ε, θα αφιερωθούν στην ε, ευέλικτη υποστήριξη στην περίοδο 2020-2021-2022 στον τομέα της υγείας, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους και σε φιλοπεριβαλλοντικά και ψηφιακά σχέδια. Και αυτά τα δισεκατομμύρια θα προσθεθούν στο τρέχον και το μελλοντικό πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και θα αποτελέσουν τη γέφυρα μεταξύ των δύο περίοδων προγραμματισμού. Το άλλο εργαλείο, το δίκτυο, το Ταμείο Δίκαιη ε, μετάβαση, ε, που είναι προσφυλέ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσφέρει 40 δι ε, εκατομμύρια ευρώ για τον κόσμο και τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τη μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερη προ τον άνθρακα. Επίσης προτείνουμε 10 δισεκατομμύριο μεσοπρόθεσμο συμπληρωματικό ποσό μέχρι το 2024 για να αντιμετωπίσουμε τι μακροπρόθεσμε επιπτώσει τη κρίση σε περιφερειακό επίπεδο στην πολιτική συνοχή το 2021 με 2027 θα πρέπει να υλοποιήσουμε τους στόχους της συνθήκη για τη σύγκληση, για τη στήριξη των λιγότερων αναπτυγμένων περιοχών της Ευρώπης και έχουμε καθήκον να εφαρμόσουμε τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες παντού, σε κάθε περιοχή, για να εξασφαλίσουμε την φιλοπεριβαλλοντική και ψηφιακή μετάβαση που δεν θα αφήνει κανέναν ουραγό. Επίσης, αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο με ένα σταθερό χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Γι' αυτό θα πρέπει το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, την επόμενη εβδομάδα να λάβει μία απόφαση και θέλουμε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμέσω μετά τη συμφωνία του Συμβουλίου. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να συνεργαστώ μαζί σα, με τα κράτη-μέλη, με τι περιφέρειε, με την κοινωνία των πολιτών, για να καταλήξουμε σε συμφωνία επί των πολλαπλών προτάσεων για τη συνοχή που έχουμε επιτάπητο. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η πολιτική συνοχή να συνεχίσει να προσφέρει έργο σήμερα, αύριο και μακροπρόθεσμα. Ε, ε, των περιφερειών και των πολιτών για μια ανθεκτική και ισχυρότερη ανάκαμψη. Είναι προς το συμφέρον μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ και προσβλέπω στη συζήτηση και στη συνεχή μας συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, κύριε Ελίζα Φεχέρα. Σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις που δώσατε στην προφορική ερώτηση. Και περνάμε στη συζήτηση με τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Η πρώτη, Μίρτσα Τζόρτζα Χάβα. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου μιλητής δυστυχώς. Micro. The micro, yes. It's okay. Okay. Again. Domnule președinte, Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η κυρία Μέρκελ, η καγκελάριος, είπε ότι θα πρέπει να φροντίσουμε τη συνοχή της Ευρώπης, γιατί είναι ουσιαστική προτεραιότητα της Γερμανικής Προεδρίας. Για να διατηρήσουμε και να εδραιώσουμε τη συνοχή μας, αυτό που χρειαζόμαστε είναι ενίσχυση της πολιτικής συνοχής, που είναι η σημαντικότερη πολιτική. Αλλιώς Πολύ σύντομα θα μιλούμε για πολιτική διάβρωση και όχι για πολιτική συνοχή. Το κείμενο αναφοράς για την Ευρώπη είναι ε, τώρα να έχουμε μεγαλύτερη υγεία, υγεία εμείς και οι οικονομίες μας αν δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα την υγειονομική κρίση και τα οικονομικά προβλήματα με αλληλεγγύη, τότε πότε θα δείξουμε αλληλεγγύη. Οι Ευρωπαίοι πολίτε χρειάζονται τα χρήματα από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και από το σχέδιο ανάκαμψη. Μπορεί να ε, είμαστε μακριά και να κρατάμε αποστάσεις, αλλά δεν ξεχνάμε ότι χρειαζόμαστε την οικονομική ενίσχυση. Τα κράτη-μέλη χρειάζονται μεταβατική ενίσχυση με σαφείς όρους για να μπορούν να απορροφήσουν ε, ε, τα διάφορα χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο οικονομικές δεσμεύσεις στα χαρτιά χωρίς ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τώρα χρειάζεται να αποφασιστεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Σας ευχαριστώ. Η Μόνικα Κονσάλες ακολουθεί για ένα λεπτό εκ μέρους των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Πολύ σαφέ το μήνυμά σα. Η πολιτική συνοχή δεν είναι θέμα αλληλεγγύη, είναι θέμα δικαιοσύνη. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλο το δυναμικό που έχουν οι περιφέρειε και οι δήμοι μα για να ε, ανοικοδομηθούμε μετά από αυτή την τρομερή πανδημία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον. Το είπατε, κατά τη διάρκεια τη πανδημία πάνω από 37 δις κινητοποιήσαμε για την ε, ε, εργασία και για όσους το είχαν ανάγκη. Ε, άτομα με αναπηρίες, άστεγοι, ηλικιωμένοι σε πόλη και σε ύπηθρο. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε που είναι κοντά στους πολίτες και όχι υπέρ των φορολογικών παραδείσων. Χρειαζόμαστε να ανακάμψει η Ευρώπη Γι' αυτό η περίοδος 21-27 και η συνοχή θα πρέπει να ε, γίνουν με επενδύσεις, όχι εκείνες που να συνδέονται με την COVID, να μειωθούν ε, οι ανισότητες και να έχουν προτεραιότητα οι δήμοι και οι κοινότητες χωρίς αιρεσιμότητα και χωρίς να μένει κανένας πίσω. Γι' αυτό ε, έχουμε να αποθέσει μεγάλες ελπίδες στο Συμβούλιο να πάρουν απόφαση για να μην ξεχάσουν κανένα και να μην έρθουν κανένα στην άκρη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Κονσάλες. Ακολουθεί η Ζωζάνα Σολής Πέρες εκ μέρους ε, της ομάδας Europe. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η πανδημία δημιουργήσε ένα προηγουμένο προκλήσεις για τα, για τα θεσμικά όργανα. Ε, κατέδειξε κάποιες αδυναμίες, αλλά είμαστε υπερήφανοι για την αντίδραση της Ευρώπης. Μάλιστα, τέθηκε σε εφαρμογή το μεγαλύτερο σχέδιο ανάκαμψη ε, που είχε ποτέ υποβληθεί στην Ευρώπη, με τη συνοχή και την αλληλεγγύη στο επίκεντρό του χωρίς, ε, ε, και σε αυτή την έκτακτη ανάγκη ο, ο ρόλος της συνοχής ήταν σημαντικός και γι' αυτό και για την ανάκαμψη τα νέα κονδύλια θα είναι σημαντικά. Θα πρέπει λοιπόν ε, να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες, να φτάσουν τα κονδύλια το συντομότερο δυνατό στους πολίτες, να έχουμε την ιδέουσα ευελιξία και να καταπολεμήσουμε ή να εξαλείψουμε τη γραφειοκρατία. Με την κρίση αυτή θα πρέπει να σκεφτούμε και τον προορισμό και τη χρήση αυτών των κονδύλιων. Γιατί τα κονδύλια αυτά είναι η ευκαιρία που θα έχουν η ε, τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι, οι κοινότητε ε, για να πραγματοποιήσουν μεταρρυθμίσει ε, που θα του επιτρέψουν να κάνουν τη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιακό, φιλοπεριβαλλοντικό και αηφόρο μοντέλο. Θα πρέπει να φτάσουν τα κονδύλια αυτά στον τουρισμό, στι μικρομεσαίες επιχειρήσει, για να γίνουν πιο ανταγωνιστικέ και πιο ισχυρές. Και θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι προτεραιότητε και τι Ευρώπη θέλουμε. Θέλω μια Ευρώπη που να είναι πιο κοντά στου πολίτε, που θα επενδύει στην παιδεία για του νέου, αλλά και στην κατάρτιση όσων εργάζονται και θα πρέπει να ανακυκλωθούν. Θέλουμε να κρατήσουμε τον κόσμο στην Ήπεθρο και να κάνουμε την Ήπεθρο ελκυστική για του νέου, για τι οικογένειε. Θέλουμε μια Ευρώπη χωρί ψηφιακό χάσμα. Θέλουμε μια Ευρώπη με μια ε, ταχεία ψηφιακή διοίκηση ε, χωρί ανισότητε, χωρί ανισορροπίε, που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω. Όλα αυτά θα καταστούν δυνατά αν όλοι συνεργαστούμε για μια πολύ πιο ισχυρή πολιτική συνοχή, μια πολύ πιο φιλόδοξη και μια πολύ σύγχρονη ε, πολιτική συνοχή. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η Αλεξάνδρα Μπάσο από την Ταυτότητα και Δημοκρατία. Ένα λεπτό. Όταν μιλάμε για πολιτική κοινωνική συνοχή για το καλό των ευρωπαϊκών λαών, δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε αυτά που συνέβησαν και αυτά που συμβαίνουν όσον αφορά την οικονομική κοινωνική κρίση που δημιουργήθηκε από τον κορονοϊό. Τόσα λόγια, δηλώσεις, αλλά μέχρι τώρα λίγες πράξεις. Είναι καλύτερο να υπόσχεται κανείς λίγα και να κάνει αυτά που υπόσχεται παρά να κάνει μεγάλες ανακοινώσεις. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία και μόνο ότι ο τρόπο θα είναι δυνατόν να μειωθούν οι αποστάσεις και να υπάρξει τελικά μεγαλύτερη ισότητα. Χρειάζονται μεγαλύτερες επενδύσεις που θα μπορούν να καλύψουν τα κοινωνικά κενά και τις διαφορές σε διάφορες περιοχές, προστατεύοντας και προωθώντας τις ιδιαιτερότητες και τις τοπικές ταυτότητες και μπορούν να ευνοήσουν ένα πλησίασμα των περιοχών και συνοχή. Αυτή είναι η πρόκληση που έχει μπροστά της Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε θα μπορέσει να αντιμετωπίσει. Ελπίζω ότι τα θλιβερά μαθήματα του COVID να μας χρησιμεύσουν. Διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Συνοχή θα επιδεινωθεί μέχρι από ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Νίκλας Νίνας για ένα λεπτό, εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Επίτροπε που ήρθατε σήμερα ε, ε, στην Ολομέλεια. Τι είδαμε όλοι ότι πρέπει να λάβουμε γρήγορα μέτρα για να βοηθήσουμε τις περιφέρειες και πολύ καλά το κάναμε μέχρι σήμερα. Τώρα όμως είμαστε σε μια διαφορετική φάση και θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαδικασία για να δούμε Ποιο χρειάζεται περισσότερη βοήθεια. Χρειάζεται πρώτα αξιολόγηση των προηγούμενων μέτρων και να δούμε τι χρειάζεται να γίνει και πώς θα γίνει αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Για την αξιολόγηση. Ξέρουμε ότι 60 ε, περιφέρειες έχουν ζητήσει να αλλάξει το έσπατος. Ε, υπάρχει καμία σχέση μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιούν τα στοχευμένα μέτρα με εκείνους που χρησιμοποιούν τα μέτρα για το COVID. Ε, το έχετε μετρήσει, το έχετε υπολογίσει και όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι για το μέλλον χρειάζεται και μια στρατηγική προσέγγιση και πώς μπορούμε να την ορίσουμε αυτή και να εξασφαλίσουμε ότι στο React EU θα έχουμε αυτή τη στρατηγική με λιγότερη Ε, με μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη απλούστευση μάλλον που χρειάζεται πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Μαγκαλία Γκυλάρ. Για ένα λεπτό, εκ μέρους των μεταρρυθμιστών συντηρητικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες ε, της πανδημίας COVID-19 είναι ολέθριες και δραματικές, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η πατρίδα μου η Ισπανία, όπου η κακή διαχείριση πολλαπλασίασε το ολέθριο αποτέλεσμα της πανδημίας. Στην ευρωπαϊκή ανταπόκριση της κρίσης, τα ταμεία και κονδύλια συνοχής έχουν ε, ζωτική σημασία για την εξάλληψη των ε, ανισοτήτων και την οικονομική ανάκαμψη που θα είναι μακροχρόνια και περίπλοκη. Ε, χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την άποψή μα και την εστερνίζεται ότι δηλαδή τα κράτη-μέλη θα μπορούν να μεταφέρουν κονδύλια μεταξύ των προγραμμάτων. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δύο εκκρεμότητε. Σε ό,τι αφορά την ε, συνοχή και την απλούστευση των διαφόρων μηχανισμών, το Ταμείο Μετάβαση δεν μπορεί να αντικαθιστά τα κονδύλια τη συνοχή, αλλά να τα συμπληρώνει σε πολύ συγκεκριμένε ε, πτυχέ. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό όπως ε, είπαν επαρελειμμένως οι προλαλήσαντες. Ε, μια φιλόδοξη ε, πολιτική συνοχή, που είναι σημαντικότερη από ποτέ σήμερα, δεν χρειάζεται περίκοπες, αλλά ένα προπολογισμό στο ύψο των περιστάσεων και των αναγκών. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό επίσης, το λόγο έχει ο συνάδελφος Ζωάν Φεχέιρα από την QNGL. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χρήση των διαρθρωτικών και επενδυτικών κονδύλιων. Έχουμε όμω ελάχιστα κονδύλια και μερικές φορές έχουμε και μεταφορά κονδύλιων από προγράμματα που τα χρειάζονταν. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι συνεχίζει να ε, επιβαρύνει τη συνοχή αφαιρώντας κονδύλια από τον προπολογισμό. Έχουμε σύμμετρα αποτελέσματα από το Σύμφωνο Σταθερότητας και και ε, το ενιαίο νόμισμα. Οπότε ουσιαστικά δεν έχουμε περισσότερη σύγκληση, αλλά όλο και μεγαλύτερη απόκληση. Επίση, μιλήσατε για το Ταμείο Συνεργασία, αλλά ευθελή είναι τα ποσά, πενιχρά. Επίση, ε, έχουμε μεταφορέ ανεξέλεγκτε και δεν θα αλλάξουμε την πραγματικότητα τη απόκληση και των διαφορών. Θα την επιδεινώσουμε. Θέλουμε περισσότερη και όχι λιγότερη συνοχή, περισσότερη και όχι λιγότερα διαρθρωτικά κονδύλια, περισσότερη υποστήριξη του παραγωγικού τομέα, του περιβάλλοντο, των επιχειρήσεων. Θέλουμε ε, περισσότερη και όχι λιγότερη ευελιξία για τη μεταφορά και επίσης ε, θα πρέπει να αυξήσουμε και όχι να περικόψουμε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και επίσης να εξελίψουμε μονίμως ε, περιορισμούς όπως του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό είναι το ελάχιστο απαραίτητο και θα πρέπει να αποκληθούν από τον υπολογισμό τα κονδύλια της συνοχής. Επίσης θέλουμε μία διάσταση συνοχής στα κεντρικά προγράμματα διαχείρισης, σε όλα τα προγράμματα, στην επιστήμη, στο περιβάλλον, και σε άλλους κλάδους και θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια ε, λογική επιμερισμένης διαχείρισης. Υπάρχουν λύσεις, αλλά δυστυχώς φαίνεται να διαφορεί για αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο Αντώνη Κομίνη Ολιβέρες για ένα λεπτό από τους μη εγγεγραμμένους. Λείπουν ακόμα τα στοιχεία, αλλά η εμπειρία μα λέει ότι μια οικονομική κρίση όπω η παρούσα θα αυξήσει τι μεγάλε οικονομικέ ανισότητε μεταξύ των πολιτών. Αυτό συνέβη μια κρίση το 2008. Δεν έχει σημασία αν οι χρηματοστικέ αγορέ είναι ένα ιό ε, οι πιο αδύναμοι πλήττονται. Στόχο τη πολιτική συνοχής είναι η σύγκληση οικονομική και κοινωνική στι ε, περιοχέ της Ένωσης. Αλλά σε μια περίοδο κρίσης αυτή ε, η, η σύγκληση σταματά. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε το διοτικό Ταμείο και τις διάφορες αρχές σε κάθε πλαίσιο. Όταν τα έσοδα τα φορολογικά των κρατών μελών ε, μειώνονται δραστικά, πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους ε, πόρους με, μέσω της χρηματοδότησης ε, όπως όταν είμαστε σε μια περίοδο ανάκαμψης. Ναι, χρειάζεται μεγαλύτερη ανα, ε, απλούστευση και ευελιξία. Δεν θα πρέπει να πάνε στους σκοπούς αυτά τα ταμεία ή θα πρέπει να εξαιρεθούν από το, το σύμφωνο σταθερότητα. Χρειάζεται πολιτική συνοχή και θα πρέπει να βγουν στο κατάλληλο πλαίσιο το παρόν τη κρίση για να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τι οικονομικέ ανισορροπίε που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των δημοκρατιών μα. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περάμε στο δεύτερο γύρο από το ΕΛΚ, ο κύριος Φρανκ Μπόγκοβιτς. Για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με, χωρίς επιτυχή πολιτική συνοχής, η Ευρώπη θα ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Θα υπήρχαν περισσότερες διαφορές. Θα υπήρχαν λιγότεροι άνθρωποι στην Ήπεθρο και δεν θα είχαν όλες τις αναγκαίες υποδομές. Η κρίση του κορονοϊού κατέδειξε ότι είναι πολύ καλή, καλό να είναι κανείς στην Ήπεθρο με καθαρό αέρα, με τον κήπο του, με ένα ροσπιτάκι. Ίσως είναι καλύτερο να ζει κανείς εκεί παρά στην πόλη. Είναι πολύ εύκολο να είναι εκεί κανείς υγιής και ε, διανοητικά υγιής στην Ήπεθρο από την πόλη. Γι' αυτό χρειάζεται κατάλληλη υποδομή. Χρειάζονται ευρυζωνικές υπηρεσίες διαδικτύου στην Ήπεθρο. Τώρα μόνο ε, οι μισοί άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο. Και αυτές ε, οι συνδέσεις θα επιτρέπουν ψηφιακή εκμάθηση, εξαποστάσεως, εκμάθηση, αγορές αποστάσεως. Όλα αυτά χρειάζονται. Και στο μέλλον η Ευρώπη ελπίζουμε ότι θα, θα χρησιμοποιήσει μέσω επενδύσεων ε, σωστά προγράμματα, να δημιουργήσουμε ευφυή χωριά, να αναπτύξουμε την Ήπεθρο και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια πράσινη και βιώσιμη Ευρώπη στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους των Συλλιστών και Δημοκρατών, Χάνες Χάιντε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η περιφερειακή πολιτική είναι η διακαριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο πολιτισμός και η παιδεία κανονικά θα έπρεπε μέσω της πολιτικής αυτής ε, ο κόσμος ε, γνωρίζει και νιώθει την Ευρώπη ε, στις πόλεις και τα χωριά. Ε, το τρίτο και πλέον των θέσεων εργασίας στην τελευταία προγραμματική περίοδο δημιουργήθηκαν χάρη στην περιφερειακή πολιτική. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες και χωρίς δεσμευμένη και φιλόδοξη πολιτική για τις περιφέρειες δεν γίνεται να τα βγάλουμε πέρα. Ε, είναι νέες οι ανάγκες και οι απαιτήσει και χρειάζονται την απαραίτητη χρηματοδότηση. Σε ένα φιλόδοξο προπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει τα περιφερειακά ταμεία να γνωρίσουν μεγάλη ενίσχυση. Μόνο έτσι τα σημαντικά θέματα του μέλλοντο, όπω η ψηφιοποίηση, η προστασία του κλίματο και η αντιμετώπιση τη κρίση θα γίνουν πραγματικότητα. Είναι θέμα αλληλεγγύης αλλά κυρίων λογική, γιατί η ωφέλεια είναι ορατή για όλους. Όσο καλύτερη είναι η περιφερειακή πολιτική και ενίσχυσή της, τόσο περισσότερο αυξάνεται η οικονομία, η εξοπιστία της Ένωσης, θέσεις εργασίας και το κοινό μας μέλλον σε μια ε, ενωμένη Ευρώπη. Των ανθρώπων όμως. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Στεφάν Μπιζού από το Renew Europe. Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Επίτροπε, σήμερα το πρωί, αυτή τη στιγμή, μία από τις περιοχές που επλήγει περισσότερο από τον κορονοϊό είναι γαλλική, στη, γαλλική Γουιάννα. Υπερπότη διαμέρισμα, η Ευρωπαϊκή Γουιάννα αντιμετωπίζει μια φρικτή υγειονομική κρίση. Ο Υπουργός ε, ο Πρωθυπουργό σε 48 ώρε θα πάνε εκεί και ο Υπουργό Υγεία για να βοηθήσουν τον πληθυσμό. Θα πρέπει να παρέμβει και η Ευρώπη. Προφανώς υπάρχει ο μηχανισμός Rescue EU, προφανώς θα πρέπει να παρέμβει. Χρειάζεται επίσης να συνοδεύσουμε τις διάφορες λύσεις, τις τοπικές, μέσω των τοπικών αρχών που χρειάζονται βοήθεια και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την επιτόπια τεχνογνωσία, αν να κάνουμε τα πάντα και να πολεμήσουμε τον ιό. Θα πρέπει επίσης όμως να πολεμήσουμε κατά του αισθήματο εγκατάλειψης έναντι του κορονοϊού που αισθάνονται εκεί. Χρειάζεται αλληλεγγύη στην Ευρώπη και η λύση υπάρχει, την έχουμε, είναι η συνοχή. Η συνοχή μεταξύ των διαφόρων περιοχών, η συνοχή μεταξύ όλων των Ευρωπαίων. Λοιπόν, η ευελιξία, η απλούστευση, η δυνατότητα αντίδραση, όλα αυτά τα εργαλεία διαχειρίσεω των κρίσεων θα πρέπει να ενοποιηθούν και να γίνουν ο κανόνα, ο κανόνας του οικοδόμησης μιας ελληλέγγυας και χρήσιμης Ευρώπης. Ευχαριστώ. Από το ECR, Ρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φέτος στην Άνοιξη το εργοστάσιο ελαστικών από του Φρέντεστάιν στο ένσεντε της Ολλανδίας ανακοίνωσε μαζικές απολύσεις. 750 ανθρώπους απέλησαν. Μετά από 110 χρόνια μετεγκαθίστανται στην Ουγγαρία όπου το 2017 το Φρέντεστάιν εγγενίασε ένα σύγχρονο εργοστάσιο. Πριν από 15 μέρες καταλάβαμε ότι πήραν χρήματα ε, στην Ουγγαρία από το Ταμείο Συνοχής για να φτιάξουν τον αυτοκινητόδρομο M3 γύρω από το εργοστάσιο αυτό. Αλλιώ δεν θα είχε φύγει ποτέ από την Ολλανδία. Χρησιμοποιούνται τώρα λοιπόν κονδύλια τη Ένωση για να προσελκύσουν εταιρείε. Ε, τι θα γίνει τώρα αν το Ταμείο Ανάκαμψη εγκριθεί των 750 δι. Σύμφωνα με τα σχέδια που έχετε 31 δις θα δώσει η Ολλανδία 4.000 ανά νοικοκυριό ε, και η Ουγγαρία παίρνει περισσότερα κονδύλια. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας ζητάνε να είμαστε αλληλέγγυοι, δηλαδή να είμαστε ένα ATM η Ολλανδία. Ε, τώρα όμως οι Ολλανδοί χρηματοδοτούν την ίδια τους τη καταστροφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποια αλληλεγγύη δείχνει απέναντι στην Ολλανδία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος και τώρα το λόγο έχει... Το λόγο έχει η ε, ε, κυρία Σμιτ Πάουερ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε, ως πρώην δήμαρχος γνωρίζω τι συμβαίνει καθημερινά και τι κάνουν οι περιφέρειες και οι δήμοι με μεγάλο πάθος, αγάπη ε, αγωνίζονται ε, να δημιουργήσουν ε, τις προϋποθέσεις για να μην φεύγει ο κόσμος. Αλλά χρειάζονται υποστήριξη το νομικό πλαίσιο και τα οικονομικά μέσα. Γι' αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί δεν είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε προτάσεις για μια μεταβατική περίοδο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε καμιά περιφέρεια πίσω στην Ευρώπη. Γιατί εκεί το πάμε εάν δεν δράσουμε. Επιτέλους, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, άρση γραφειοκρατίας και θα πρέπει με αποφασιστικότητα να τα λύσουμε. Ε, ευελιξία, ελαστικοποίηση με το, τη χρηματοδότηση κατά του κορονοϊού βοήθησαν, αλλά δεν μπορούν παρά να είναι μόνο η αρχή. Γι' αυτό φροντίστε με γρήγορη δράση περιφέρειες της Ευρώπης, η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας μας, ε, να, να μην ε, αφαιθούν στη μοίρα τους μόνο με κούφια λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στην Κριστίνα Μαέστρε Μαρτίν Δε Αλμάγρο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, πριν από λίγους μήνες, όταν δεν γνωρίζαμε καν την ύπαρξη του COVID, συζητούσαμε εδώ για την ε, πιθανότητα ενός πιο φιλόδοξου πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου και δεν μας άρεσε η απειλή περικοπής των κονδυλίων της συνοχής και ζητήσαμε λιγότερη ανελαστικότητα και περισσότερη ευελιξία. Φαίνεται ήταν χήμερα αυτή η φιλοδοξία μας. Βέβαια, φάνηκε από την πανδημία ότι όταν ε, θέλει κανείς μπορεί να το επιτύχει κάτι. Χρειάζεται απλώς βούληση. Τώρα, δυστυχώς, ε, εμ, δόθηκαν κάποια βοήθεια, αλλά θα πρέπει να μείνουμε στην ε, Στι πρώτε βοήθειε που παρίσχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε χωρί αιρεσιμότητα να δώσουμε κονδύλια για να μην απο... επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Πώ θα το καταφέρουμε. Επίση, τι θα ακολουθήσει η πολιτική συνοχή ε, είναι ο ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού οικοδομήματο, του ευρωπαϊκού σχεδίου. Δεν μπορούμε αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο να τον ε, πλήξουμε ή να τον αφήσουμε να καταρρεύσει από την κρίση. Αντίθετα από την κρίση, θα πρέπει να τον ενισχύσουμε, να δώσουμε και ποσοτικά και ποιοτικά το ρόλο που αξίζει στην πολιτική συνοχή. Και μπορείτε να υπολογίζετε στη δική μα συνδρομή για να το επιτύχουμε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Ιζαμπέλ Μπεχουμέα Μπεχουμέα για ένα λεπτό εκ μέρου του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επίτροπο Φεραίρα και να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Μαρτζή που υπέβαλε την προφορική ερώτηση και μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε το τόσο σημαντικό θέμα του ρόλου των κονδυλίων της συνοχής στη διαδικασία της ανάκαμψης και της αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19 και των συνεπειών της. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή αντέδρασαν άμεσα και έγκαιρα. Είναι σημαντικό αυτό να το επισημάνουμε και στου Ευρωπαίου πολίτε. Επίση, χαιρετίζω το φιλόδοξο σχέδιο που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Next Generation EU. Μιλάμε για 750 δισεκατομμύρια ευρώ που θα προέλθουν από, τα, ε, από τους φόρους των Ευρωπαίων πολιτών και θα τροφοδοτήσουν την πολιτική συνοχής για την εποχή μετά την επιδημία, την πανδημία COVID είναι σημαντικό τα κονδύλια αυτά να χρησιμοποιηθούν στις περιοχές που πληγήσαν περισσότερο από τις επιπτώσεις της κρίσης COVID-19. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τα κονδύλια να δρομολογηθούν προς τις πληγήσεις περιοχές κυρίως. Επίσης, να κάνουμε μια επανειεράρχηση των προτεραιοτήτων και να έχουμε ως υπέρτερο στόχο τη δημιουργία πλούτου και απασχόλησης και να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ας μην ξεχνούμε λοιπόν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να υποφεληθούν κυρίως από τα κονδύλια της συνοχής και που θα εγκριθούν ε, στο πρόγραμμα Next Generation EU, στο σχέδιο δηλαδή της ανάκαμψης. Ευχαριστώ. Και τώρα για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση θα ξαναδώσω το λόγο στην Επίτροπο Φεχαίρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη που μας προσφέρατε, που δώσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πολλές φάσεις και στις δύσκολες στιγμές που περάσαμε. Θα ήθελα πρώτα να αναφέρω αυτό που είπε ο κύριος Χάιντε, ότι η πολιτική συνοχής είναι η παλόμενη καρδιά της Ευρώπης. Το πιστεύω αυτό και παλόταν ακόμη και σε δύσκολους καιρούς, ακόμη και όταν είχαμε προβλήματα, ακόμη και όταν υποφέραμε. Και σας ευχαριστώ κύριε Ομαρζή που αναφερθήκατε στο έργο που επιτελέσαμε από κοινού και προσφέραμε άμεση αντίδραση για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία COVID-19. Επίσης, αυτή η ευκαιρία που ανέφεραν οι συνάδελφοι ότι, ότι υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένε καταστάσει, να φτάσουν αυτά τα κονδύλια στον κόσμο, στι περιοχέ και η ελαστικότητα που προβλέπουμε, η ευελιξία που προβλέπουμε στην αντίδραση του κρί και κρίσιν ε, νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Μέχρι στιγμής όλα τα κράτη-μέλη, με εξαίρεση την Αυστρία και τη Δανία, χρησιμοποίησαν τις δυνατότητες μεταφορών για τη χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων. Και μιλάμε για πάνω από 50 δις το πολύ για να πληρώσουν τα κράτη-μέλη ε, τις χειρουργικές μάσκες, τις αναπνευστήρες, να στηρίξουν τις θέσεις απασχόλησης, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δώσουν μια άμεση απάντηση να ανταποκριθούν άμεσα. Είπατε ότι η πολιτική συνοχή είναι η παλιά πολιτική και όμως είναι ζωντανή, ακμαία και μπορεί να παράσχει την έκτακτη βοήθεια όταν χρειάζεται. Βέβαια, ε, δεν είναι η μόνη χρηματοδοτική πολιτική αυτή η πολιτική συνοχή, αλλά είναι η μεγαλύτερη και η πιο ορατή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, ως προς την ποιότητα των προτάσεών μας, χρειάστηκε να προτείνουμε ε, μακροπρόθεσμες δράσεις που θα συνδυάζουν όμως και βραχυπρόθεσμους μηχανισμούς όπως το React-EU και θέλουμε να κρατήσουμε ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και να υπάρχει δυνατότητα ε, χρηματοδότηση έως και 100% αν το αποφασίσουν τα κράτη-μέλη. Βέβαια το react e για πρακτικούς λόγους δεν μπορεί να διανεμηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθείας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Γιατί εμείς ε, κατανέμουμε τα κονδύλια με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία. Μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού δεν θα έχουμε ακόμη τα στοιχεία από περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη όμως θα μεταφέρουν τα ίδια κριτήρια που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή τη μείωση του ΑΕΠ, τη μείωση της ανάπτυξης, αύξηση της ανεργίας, της ανεργίας των νέων. Όλα αυτά τα κριτήρια θα ληφθούν υπόψη. Επίσης, η σχετική ευημερία της χώρας είναι ένα κριτήριο που θα ληφθεί υπόψη για να δημιουργηθεί μια γέφυρα με το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μια γέφυρα που θα βοηθήσει τις περιφέρειες να μειώσουν τις διαφορές τους. Επίσης, ε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη την ποιότητα και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη σε αυτή την κατανομή των κονδυλίων. Και εδώ προσπαθώ να απαντήσω ε, και στην ερώτηση του κυρίου Μαρζή. Επίσης, ε, θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Ναι, είναι σημαντικό να λάβουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως τη βάση και θα πρέπει να σταματήσουμε να λέμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια. Υπάρχουν αρκετά χρήματα. Κύριε Νίνας, είπατε και κάποιοι άλλοι νομίζω το ανέφεραν, είπατε ότι θα πρέπει να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε με αυτά τα χρήματα και θα πρέπει να είναι ποιοτική η ανταπόκρισή μας, γιατί η ποιότητα των δράσεών μας θα επηρεάσει το μέλλον μας. Και τώρα, σε σχέση με τα, σχόλια, του κυρίου Φερέρα που είπε ότι ίσως ε, καταρρεύσουν κάποια ταμεία. Όχι, δεν θα υπάρξει έλλειψη κονδυλίων. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα κονδύλια του ΠΔΕΛΤΑΠΗ και να τα συνδυάσουμε με τους συμπληρωματικούς μηχανισμούς που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε 55 δισεκατομμύρια ευρώ για το React-EU καταρχάς. Επίσης 32,5 δισεκατομμύρια για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και 10 δισεκατομμύρια ευρώ ε, που θα έρθουν ε, συμπληρωματικά στο 2020 και θα καταμεριστούν ανάλογα με τα κριτήρια της αύξησης ανεργίας και μείωση της ε, ανάπτυξης στα διάφορα μέρη της Ευρώπης. Πάνω από 100 δισεκατομμύρια δηλαδή συνολικά. Και αυτό που προέχει είναι το συντομότερο δυνατό να, να διαμορφώσουμε μια σαφή εικόνα και ικανότητα για να οργανώσουμε τις δράσεις μας και να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε εμπράκτος και σωστά όλες αυτές τις ευκαιρίες που δημιουργούμε. Πάντως είμαι πολύ περήφανη που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν τόσο τολμηρή ε, και τόσο φιλόδοξη στις προτάσεις της. Και αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην πίεση που άσκησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, δόθηκε ε, όθηση και από διάφορες κυβερνήσεις ε, και καταφέραμε και αναλάβαμε δράση. Θα πρέπει να το συνεχίσουμε και θα πρέπει ε, μετά την έγκριση να τελειοποιήσουμε κάποια σημεία, να τα βελτιώσουμε, αλλά να κινηθούμε το συντομότερο δυνατό γιατί τα κονδύλια υπάρχουν και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια συνέχεια, να μην υπάρχουν διακοπές, να εξασφαλιστεί μια συνέχεια και να λάβουμε υπόψη την ψηφιακή μετάβαση, τη σύγχρονη μετάβαση, τη φιλοπεριβαλλοντική μετάβαση που δεν θα αφήνει κανένα πολίτη πίσω, καμία περιοχή πίσω. Δεν θα πρέπει να έχουμε αποκλεισμού. Αυτές οι προτάσεις έχουμε επιτάπητος. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε τα θεσμικά όργανα για να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών σε αυτές τις κρίσιμες και δύσκολες στιγμές της ιστορίας της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ και συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Και φυσικά έχουμε κυρίως κατά νου τις ε, περιοχές με τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Ε, ήμασταν ανέκαθεν ε, υπέρ αυτών των περιοχών και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί θα πρέπει όλοι να συμμετέχουν σε αυτό το κοινό μας μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Προεπίτροπε και για την παρέμβασή σας και για το έργο σας. Δεν έχουμε κάθε μέρα επίτροπο να μας λέει λεφτά υπάρχουν και πολλά μάλιστα. Σπάνια ακούμε κάτι τέτοιο. Περιμένουμε φυσικά τι αποφάσει του Συμβουλίου και α μην ξεχνούμε ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει τον τελικό λόγο, την τελευταία λέξη ε, και θα διατρανώσει τη θέση του υπέρ της πολιτικής συνοχής. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για τη συμμετοχή σας. Ολοκληρώνεται η συζήτηση και του αυτού και διακόπτουμε τις εργασίες της Συνόδου της Ολομέλειας μέχρι τη 1.30.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

1, 2, 3, 4. okay. So, good afternoon, colleague. Καλησπέρα συνάδελφοι. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση και τώρα θα ανακοινώσω τα αποτελέσματα της πρώτης ε, ε, συνεδρίασης ψηφοφοριών. Έκθεση κούσμα για τις ε, πολιτικές απασχόλησεις εγκρίνεται. Η έκθεση της κυρίας Χόλμαϊερ για το διορθωτικό προπολογισμό υπαρθμών 5 εγκρίνεται. Η έκθεση της κυρίας Χόλμαϊερ για την κινητοποίηση του περιθωρίου ασφαλείας επίσης εγκρίνεται. Το ψήφισμα της Επιτροπής ΕΜΒΗ για το τριοξίδιο χρωμίου απορρίπτεται. Το ψήφισμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος για τις δραστικές ουσίες εγκρίνεται. Η έκθεση της κυρίας Γκάμον για την αποθήκευση ενέργειας εγκρίνεται. Το ψήφισμα της Επιτροπής Ήτρε για τις υποδομές TEN-E ε, εγκρίνεται. Προχωράμε στην τροποποίηση του κανονισμού 2016 κάθετος 1628 που αφορά τις, μάλλον όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της κρίσης COVID-19. Τροπολογία 4 πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Τροπολογία 3 απορρίπτεται. Τροπολογία 1 απορρίπτεται. Τροπολογία 2 απορρίπτεται. Τροπολογία 4, δεύτερο τμήμα, εγκρίνεται. Προχωράμε τώρα στο αποτελέσματα της ψηφοφορίας όσον αφορά τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών. Τροπολογία 1 απορρίφθηκε. Τροπολογία 2 απορρίφθηκε. Τροπολογία 3 απορρίφθηκε. Τροπολογία 5 απορρίφθηκε. Τροπολογία 6 απορρίφθηκε και η τροπολογία 4 απορρίφθηκε. Αναστολή, διακοπή μάλλον, μέχρι τις 14 και 15.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 Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Παρακολουθείτε την Ολομέλεια κατά πάσα πιθανότητα από τα γραφεία σας. Είμαστε στον δεύτερο κύκλο ψηφοφορίας για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και είναι από τώρα 2,5 μέχρι τις 3,5. Αρχίζει λοιπόν η δεύτερη ψηφοφορία και έχετε μέχρι τις 15 και 30 για να ψηφίσετε και στις 6 το απόγευμα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Έχω και κάποιες... Δεν έχω μάλλον άλλες ανακοινώσεις. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. μετά. Ε, εντάξει. Ναι, Presidente. So. η συνεδρίαση. Θα σας ανακοινώσω τα αποτελέσματα της δεύτερης ψηφοφορία. Καταρχάς, ό,τι αφορά την έκθεση σύναψη τη υποδιαπραγμάτευση Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Νέα Ζηλανδία σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματο και τη τρομοκρατία εγκρίνεται. Είχαμε ε, για την ε, ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος Έκθεση για τη Στρατηγική και τις Χημικές Ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα εγκρίνεται. Έπειτα είχαμε τις μεταβατικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της νόσου COVID-19. Εγκρίνεται. Πρώτη ανάγνωση λοιπόν του Κοινοβουλίου εδώ ολοκληρώνεται. Επίση, ό,τι αφορά τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών με φάρμακα για ανθρώπινη χρήση, περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού και τα οποία προορίζονται για τη θεραπεία, την πρόληψη τη από κορονοϊό και προμήθεια τέτοιων φαρμάκων με την κατεπίδουσα διαδικασία. εγκρίνεται και ολοκληρώνεται και για αυτήν ε, την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Έπειτα έχουμε από πέντε ομάδες ε, μια κοινή πρόταση ψηφίσματο για μια ολοκληρωμένη πολιτική τη Ένωση για την πρόληψη τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε και τη χρηματοδότηση τρομοκρατία. Εγκρίνεται και αντικαθιστά τις άλλες εγκρίνεται και η σχετική έκθεση. Και έπειτα έχουμε την κοινή πρόταση ψηφίσματο για τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Δημόσια Υγεία μετά την κρίση COVID-19. Εγκρίνεται. Θέλω επίσης να σας πω ότι είχε υπογράψει δύο νομοθετικέ ε, πράξει ε, μετά τη διακοπή τη Συνόδου περίοδου 19η Ιουνίου, ο πρόεδρο του Κοινοβουλίου μαζί με τον πρόεδρο του Σύμβουλου Δυνάμει του άρθρου 79 και μετά τις 15 Ιουλίου οκτώ νομικές πράξεις θα καταγραφούν στα πρακτικά οι νομοθετικές αυτές πράξεις σε ό,τι αφορά των τίτλων του ε, Επίσης 8, 9, και 10 ε, Ιουλίου. Ε, έχουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων που αν δεν υπάρξει κάποια ένσταση θα εγκριθούν στην έναρξη της επόμενης συνόδου όλο μέλη. Θα τεθούν για έγκριση. Αν δεν υπάρχουν ε, ενστάσεις θα διαβιβάσω στους αρμοδίους αυτά τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στην τρέχουσα ολομέλεια. Εδώ θα ολοκληρωθεί η Σύνοδος Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο πέρα στη συνεδρίαση. So, I take the free drink.